Συνάδελφοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στη συνεδρία της Επιτροπής μας και να καλωσορίσω και τον πρώτο αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Φραντ Τιμερμάν, ο οποίος θα μας απευθυνθεί εντός ολίγου. Να ξεκινήσουμε με το σημείο 1 έγκριση της ημερήσιας διάταξης, να σας ενημερώσω ότι τα σημεία 12 και 13 θα εξεταστούν μετά τις αυριανές ψηφοφορίες και όχι σήμερα. Αυτή είναι η μόνη αλλαγή που προτείνεται στην ατζέντα. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Νομίζω πως όχι, οπότε θεωρούμε εγκεκριμένη την ημερήσια διάταξη. Ως προς το σημείο 2, ανακοινώσω του πρόέδρο δεν έχω τίποτε να ανακοινώσω. Σημείο 3 έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσει ω το τέλο αυτή τη συνεδρίαση, τα, τα πρακτικά θα θεωρηθούν εγκεκριμένα. 12 και 11 Απριλίου 2017 και 3 και 4 Μαΐου 2017. Οπότε μπορούμε να περάσουμε απευθείας στο σημείο 4. Ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Φρανς Τίμερμανς, στον οποίο δίνω τον λόγο ευθύς αμέσως. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι μεγάλη μου χαρά που μπορώ να είμαι πάλι στην Επιτροπή σας, που είναι και δική μου. Γιατί πολλά από τα ζητήματα που απασχολούν εμένα πρέπει να τα δω από κοινού μαζί σας. Να περιγράψω λίγο το πλαίσιο εντό του οποίο συζητούμε. Σήμερα ξεκινήσανε και πραγματεύσει για τον Brexit Στην ουσία ενημερωθήκαμε για το τι θέλουν οι Βρετανοί και τι περιμένουν. Επίσης υπάρχουν εξωτερικές εξελίξεις. Ο Πούτιν δεν αλλάζει τη γραμμή του. Ο Τραμπ είναι μια επιπλέον δυσκολία καθώς αποσύρθηκε από τη Συμφωνία των Παρισίων. Η μετανάστευση συνεχίζει να είναι ένα πρόβλημα. Είχαμε έτη όπου Όλες αυτές οι τάσεις, όλες αυτές ε, οι κινήσεις, οι εξελίξεις δημιούργησαν κεντρόφυγες τάσεις ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυγόκεντρες μάλλον. Ε, εδώ βλέπω να υπάρχει μια διαφορετική τάση για πολύ σημαντικά ζήματα και επειδή ό,τι κάνουμε πρέπει να βασίζεται στην νομοθεσία μπορούμε να πούμε δικαιολογημένα ότι αυτή η Επιτροπή θα πρέπει να δει όλα τα επόμενα βήματα της συνεργασίας μας αλλά προτού γίνει αυτό θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι τα πάντα γίνονται σωστά βάσει των υπερχουσών συνθήκων για να αγγίξω έτσι και το θέμα της διαφάνειας. Νομίζω ότι έχουμε επικοδομητικές ε, διαπραγματεύσεις βάσει της διαθεσμικής συμφωνίας και ως προς το σημείο που αφορά το υποχρεωτικό ε, μητρό ε, διαφάνειας μπορεί, εάν θέλει το Κοινοβούλιο, να συμβληθεί. Είναι ένα μητρό που εάν κανείς δεν έχει καταγραφεί ως λόμπι, μελο λόμπι, δεν μπορεί να οργανώσει συνάντηση, η συνομιλία. Καταλαβαίνω ότι αυτό διαφέρει βέβαια στη λογική του από τα λόμπι για το Κοινοβούλιο. Δεν μιλάμε όμως για συνάντηση με ψηφοφόρους σας, μιλάμε για συνάντηση με εκπροσώπους λόμπι, ομαδών πίεσης, ομάδες συμφερόντων δηλαδή, για τα θέματα τα οποία σας απασχολούν. Και επειδή έχω υπάρξει ευρωβουλευτής πάνω από μια δεκαετία, δεν θα ήθελα κανείς να μου καθορίσει πώς θα έρχομαι σε επαφή με τους ψηφοφόρους μου, αλλά ε, είναι άλλο όταν μιλάμε για ανθρώπους που εκπροσωπούν ομάδες συμφερόντων. Εκεί πρέπει να είναι γνωστό με ποιους έρχομαι σε επαφή όταν αυτοί εκπροσωπούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Είναι σημαντικό το βάση ποιών πληροφοριών ε, ε, λαμβάνω τις αποφάσεις μου και νομοθετώ. Για την καλύτερη νομοθεσία νομίζω ότι βελτιώσουμε τον τρόπο που δουλεύουμε, ιδίω χάρη στη θεσμική συμφωνία για την καλύτερη νομοθεσία, συμφωνία που επιτέχθη μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων και υπάρχει και πλατφόρμα Refit, η οποία προχωράει καλά με αρκετές γνωμοδοτήσεις, αντιδρούμε σε όλες αυτές όπως δει. Είναι ένα μεγάλο, ένας μεγάλος φόρτος, αλλά θα συμβάλλει στην καλύτερη νομοθεσία, γιατί η καλύτερη νομοθεσία δεν σημαίνει μόνο περιορισμό του γραφειοκρατικού άχθου σημαίνει ότι η νομοθεσία εξυπηρετεί του σκοπού για του οποίου σχεδιάζεται. Και αυτό σε πολλού πολλού τομεί, παλιού και νέου, ε, δείχνει ότι η νομοθεσία χρειάζεται να βελτιωθεί. Βεβαίω υπάρχει και η επόμενη φάση τη διαθεσμική συμφωνία που πρέπει να υλοποιηθεί, δηλαδή η ανταλλαγή πληροφοριών, συνεργασία και διαπραγματεύσει και η ε, περάτωση διεθνών συμφωνιών. Ξεκινήσαμε στα τέλη τη περασμένη χρονιά στην συνάντηση ομάδα υψηλού επίπεδου και ελπίζουμε ότι η ανάλογη επόμενη συνάντηση θα γίνει τον επόμενο μήνα. Επίση, θα πρέπει να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει για να καθοριστεί η διαφορά μεταξύ των καταξουσιοδότηση και των ε, Ε, και των ε, εκτελεστικών πράξεων. Ε, εδώ θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασχοληθεί με την διαδικασία για τα θέματα που έχουν ξεκινήσει λόγω της διαδικασίας του διακανονισμού της Λισαβόνας. Βεβαίω, τα κράτη-μέλη ακόμη δεν επιλέγουν εύκολα τι κατεξουσιοδότηση πράξει, ακόμη και όταν αυτέ αρμόζουν περισσότερο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίζει να επιχειρηματολογεί υπέρ του και ελπίζουμε να στηριχθούμε εδώ και από το Κοινοβούλιο. Ένα άλλο στοιχείο που έχει σχέση με την καλύτερη νομοθεσία και την, ε, τις είναι το σχετικό αρχείο που θα πρέπει να καταρτιστεί ως το τέλος της χρονιάς. Επίσης υπάρχει και ο κανονισμός της επιτροπολογίας να βεβαιωθούμε ότι κανένας δεν μπορεί να αποποιηθεί τις πολιτικές του ευθύνες γιατί και οι πολίτε και οι επιχειρήσει χρειάζονται σαφήνεια. Έχουμε δει πολλέ περιπτώσει όπου τα εθνικά κράτη-μέλη δεν συμφωνούν εσωτερικώ και μετά πετάνε τον παλάκι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να λάβει εκείνη τι αποφάσει που δεν είναι σε θέση να λάβουν. Δεν είναι αυτή όμω η συλλογιστική όλη αυτή τη προσπάθεια. Η ευθύνη θα πρέπει να αντιλαμβάνεται και από τα κράτη-μέλη. Ναι. Επίση, η επικουρικότητα και η αναλογικότητα είναι θέματα που πρέπει να υπάρξει ανάλυση, ανάληψη ευθύνη. Απευθυνόμαστε στο Εθνικό Κοινοβούλιο και μέσω της, στα Εθνικά Κοινοβούλια και μέσω τη ΚΟΖΑΚ και με 500 επισκέψει κατά διάρκεια αυτή τη θητεία. Η αναλογικότητα και η επικουρικότητα βρίσκονται στον πυρήνα τη δουλειά μα και όπου μπορούμε να έχουμε συνεργασία μαζί σα για τα θέματα αυτά θα έχουμε. Και πριν ολοκληρώσω πολύ γρήγορα για το κράτο δικαίου, η Επιτροπή αυτή ξέρουμε ότι δίνει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό, στο επιχειρησιακό περιβάλλον, στην ε, εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς που βασίζεται πάρα πολύ στην εμπιστοσύνη, την ε, ε, ασφάλεια και τα ανεξάρτητα δικαστήρια. Όλο και περισσότερο μας ανησυχεί λοιπόν η κατάσταση στην Πολωνία και σε σχέση με το νομοσχέδιο που θα ε, συζητηθεί σύντομα, εάν θέλετε να το σχολιάσω το θέμα αυτό με τα χαράς, αλλά είναι μια πολύ δύσκολη φάση στην διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης για να έχουμε αποτελέσματα και να δούμε και ποιε είναι οι κατευθύνσεις στις οποίες οδεύουμε, αλλά για να υπάρχει και μια αίσθηση ότι υπάρχει κάποιος σκοπός σε όλα αυτά και ότι υπάρχει και πρόοδος. Μόνο μαζί με τους πολίτες μας μπορούμε να καταπολεμήσουμε μαζί τον εθνικισμό, τον λαϊκισμό και την ξενοφοβία. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν ότι θεσμικό είναι απαραίτητο, αλλά ε, στο κάτω-κάτω δεν είναι μόνο αυτό που θα αγγίξει τις καρδιές των ανθρώπων. Σήμερα η Ευρώπη παρουσιάζει μια τελείως διαφορετική εικόνα από ό,τι συνέβαινε πριν από ένα χρόνο ή δύο. Ε, έχουμε να κάνουμε συγκεκριμένε επιλογέ, μα πιέζει το Brexit, αλλά υπάρχει και μια συγκεκριμένη πραγματικότητα όπου πρέπει να διαμορφώσουμε το μέλλον μα σε αυτόν τον γρήγορα μεταβαλλόμενο κόσμο. Και τα νομικά θέματα δεν είναι απλώ εργαλεία, είναι θέματα ουσία. Γι' αυτό μιλάμε για το κράτος δικαίου και όχι απλώς το κράτος ε, που, που επιβάλλει το δίκαιο του. Γι' αυτό θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ένωση όπου το κράτος δικαίου είναι διαρκώς το θεμέλιο της δουλειάς μας και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank you very much. Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Οπότε λοιπόν, τώρα έχουμε πολύ χρόνο για ανταλλαγή απόψεων με τον πρώτο αντιπρόεδρο της ε, Κομισιόν. Η κυρία Χάνιμπολ ζήτησε τον λόγο. Ευχαριστώ που ήρθατε να μας μιλήσετε. Ε, αισθάνομαι ότι πρέπει να ζητήσω συγγνώμη που είμαστε τόσοι λίγοι εδώ. Ε, που είναι λυπηρό γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία είπατε και ως Βρετανίδα προφανώς θεωρώ πως είναι πολύ σημαντική η στιγμή για το Ηνωμένο Βασίλειο. Και μιλήσατε για εθνικισμό και ξενοφοβία και χάρηκα που τα αναφέρατε αυτά. Και η Κομισιόν κοιτάει τα πράγματα και πώς μπορούμε να μειώσουμε ε, και να εξαλείψουμε αυτά τα φοβερά πράγματα από την Ευρώπη. Μια που δεν υπάρχουν άλλοι Βρετανοί, εγώ θα πω το εξή. Ε, θεωρώ ότι αυτά τα πράγματα ήταν τμήμα του Βρετανικού δημοψηφίσματος ε, και τη εξαρτία και του τι συνέβη. Τι συνέβη. Λοιπόν, έχει περάσει ένας ε, χρόνος και είναι πολύ περίεργα τα πράγματα λόγω της προσέγγισης ε, του Ηνωμένου Βασιλείου και της ε, κυβέρνησής μας. Είπατε ότι έχετε μια ξεκάθαρη ιδέα για το πού πηγαίνετε. Δεν ξέρω αν σημαίνει το ίδιο με τη Βρετανική κυβέρνηση. Μπορείτε λοιπόν ε, να μας πείτε κάποιες σκέψεις. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πράγματα που δεν μπορείτε να πείτε, αλλά λίγο να επεκτείνετε αυτά τα οποία μας είπατε. Η κυρία Κάουφμαν. κύριε Αντιπρόεδρε της ε, Επιτροπής. Καλώς ήρθατε και από μένα. Πράγματι είναι κρίμα που έχουν έρθει τόσο λίγοι συνάδελφοι. Αλλά εντάξει. Εγώ είμαι εδώ, εσείς είστε εδώ. Και χαίρομαι για αυτά τα οποία είπατε. Πριν από 1,5 χρόνο δεν θα μπορούσα να σκεφτώ ότι θα ήμασταν στην κατάσταση που περιγράψατε. Φοβόμουν ότι το, το δημοψήφισμα θα οδηγούσε σε ένα ντόμινο. Διάβασα το ότι ζήτησε ο πρώην Τσέχος πρόεδρος μετά την διαδικασία επί παραβάση για τους πρόσφυγες ε, να φύγει η Τσεχία από την Ένωση. Δεν το αντιλαμβάνομαι. Υποτίθεται ότι είμαστε μια κοινότητα δικαίου. Και όλοι πρέπει να έχουμε τις ίδιες αξίες, ε, τις ίδιες αρχές για να αναπτύξουμε αυτή την κοινότητα. Για να υπάρχει μια κοινή εμπιστοσύνη. Μιλήσατε για ένα άλλο θέμα για τις πράξεις ε, ξέρω, Μπορείτε να κάνετε κάποιες δηλώσεις. Γνωρίζω ότι είμαστε εν το μέσο της διαδικασίας και θα συζητήσουμε αυτό το θέμα τον κύριο Σάρια. Αλλά είναι κρίμα το ότι οι διαπραγματεύσει που θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει ακόμα εκκρεμούν. Ε, Πώς αυτό οφείλεται στο ότι δεν ήταν σε θέση τα θεσμικά όργανα να καθορίσουν μια θέση. Κάτι άλλο τώρα, τελείως διαφορετικό, αλλά έχουμε ώρα. Είναι το θέμα των ε, καταγγελόντων. Θέλουμε εδώ να κάνουμε μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για μια πανευρωπαϊκή προστασία τους. Και θα θέλαμε η Κομισιόν να στηρίξει ε, και να υποβάλει κάποιες σχετικές ε, προτάσεις. Υπάρχει κάποια διαμάχη που λέει ότι προστατεύονται μόνο αν αποκαλύπτουν πράγματα από ιδιωτικές εταιρείες ή μόνο εάν αφορά το δημόσιο συμφέρον. Εμεί θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας κανόνας έτσι ώστε ανεξαρτήτως από πού προέρχονται να έχουν μια προστασία και γιατί δεν είναι δυνατόν αυτοί οι οποίοι αποκαλύπτουν διάφορες ε, τέτοιες ε, κακές πράξεις και ενημερώνουν τις αρχές να, να την πληρώνουν και από πάνω. Και να τιμωρούνται στην προσωπική του ζωή επειδή αποκάλυψαν την αλήθεια. Δεν ξέρω αν μπορείτε και εδώ να μας πείτε κάτι. Ε, Mr. Anderson. Κύριε Άντερσον, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξεκινήσω με το να συμφωνήσω στα κυριότερα σχόλια. Την ανάγκη δηλαδή προστασίας ε, των καταγγελόντων. Έχω επίσης ε, μία ερώτηση για το Brexit. Είδαμε στα ΜΜΕ ότι ο κύριος Φερχόφστατ είπε ότι μήπως πρέπει η Βρετανία να ξανασκεφτεί και αν δεν ξανασκεφτεί την απόφασή της δεν μπορεί να συνεχιστούν διαπραγματεύσεις με τους υφιστάμενους όρους αλλά με χειρότερους π.χ. όσον αφορά την επιστροφή χρημάτων. Ε, αυτή είναι η άποψη της Κομισιόν ή όχι. Επίσης, Πενιχθήκατε ότι έχετε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα να πείτε για την Πολωνία και το κράτος δικαίου. Και θα ήθελα να τα ακούσω και αυτό. Σας ευχαριστώ κύριος Λεμπρετόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να καλωσορίσω και εγώ τον κύριο Τίμερμαν. Πάντοτε είναι μια σημαντική στιγμή όταν υποδεχόμαστε στην ε, Επιτροπή μας, τον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είπατε το Μάρτιο, κύριε Τίμπερμαν, ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να δημιουργηθεί σε βάρος ε, των ε, εθνών κρατών. Μου άρεσε πάρα πολύ που το άκουσα αυτό, φαντάζομαι το καταλαβαίνετε. Ωστόσο, Νομίζω ότι τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει το αντίθετο, παρεμβαίνει δηλαδή τα μάλα στι εσωτερικέ υποθέσει ορισμένων κρατών μελών. Μιλήσατε για την Πολωνία και ουσιαστικά μα τίνατε έτσι και μια παγίδα λέγοντα να ε, μιλήσουμε πιο πολύ για αυτά. Ε, μία πολωνική εφημερίδα σας ε, έχει εκλέξει άνδρα ε, του προσωπικού του 2017. Αυτό δείχνει ότι τελικά πράγματι η Κομισιόν έχει παρέμβει σημαντικά σε εσωτερικές υποθέσεις Πολωνίας. Και αυτό που έχω καταλάβει εγώ από τα πολωνικά αυτά θέματα είναι ότι τελικά αφιζητείται ένα ε, project ε, μεταρρυθμίσεων ε, της δικαιοσύνης και νομίζω ότι αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει γιατί είναι εθνικό κυριαρχικό δικαίωμα της κάθε χώρας να αποφασίσετε της δικαιοσύνης ως κρίνη. Επίσης θα ήθελα να μας μιλήσετε για την Ουγγαρία, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει να προσάψει πολλά στην Ουγγαρία και ιδίως σε ό,τι αφορά δύο ζητήματα πολύ επίκαιρα. Το ένα αφορά την υποτιθέμενη τουλάχιστον παραβίαση της ελευθερίας εγκατάστασης. Αναφέρομαι σε ένα νομοσχέδιο που θα θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία του Πανεπιστημίου του Σόρους, αλλά αν δούμε το σχέδιο, αυτό δεν είναι και τόσο πια ριζοσπαστικό όσο ακούγεται ότι είναι, γιατί το μόνο που θα δημιουργήσει πρόβλημα είναι ε, να ξέρουν πανεπιστημίο όταν δεν έχουν αιστεία ε, στην ε, χώρα καταγωγής ε, δηλαδή ουσιαστικά πολύ λίγο αυτό αφορά το ίδιο το Πανεπιστήμιο και δεν ξέρω κατά πόσο τελικά είναι θεμητό ένα κράτος μέλος ε, να ψηφίσει τέτοιου είδου νομοσχέδια. Σας ερωτώ απλά. Και ένα άλλο νομοσχέδιο που δημιουργεί πολλά προβλήματα είναι ένα νομοσχέδιο που θα δίνει τότε δυνατότητα στις Ουγγρικές αρχές ε, πολύ εύκολα να προσάγουν μετανάστε που φτάνουν στη χώρα, του. Μπορούμε να το συζητήσουμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά και ο συστηματικό χαρακτήρα των προσαγών και των κρατήσεων. Αλλά νομίζω ότι επίση θεμητό είναι να ενδιαφέρεται και να ανησυχεί ένα κράτο μέλο για τι μεταναστευτικέ ροέ. Αυτά και περιμένουμε υπομονησία τη απαντήσει σα. Ο κύριος Φω. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Δύο ερωτήσεις έχω ή μία αφορά την συνοχή νομοθετημάτων όπου βλέπω μία ψαλίδα να ανοίγει που ίσως να μην ήταν ε, η πρόθεση αλλά αυτό συμβαίνει τελικά. Και το άλλο είναι ότι πρέπει ε, εκ των προτέρων να δούμε κάποια πράγματα ενιολογικός πώς. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Το ένα είναι έχουμε επίχει τον κανονισμό που εγκρίναμε πέρσι το Μάιο για την προστασία των δεδομένων και θα αρχίσει να ισχύει του χρόνου το Μάιο. Και έρχεται τώρα πρόταση για ηλεκτρονική ιδιωτικότητα. Εντάξει, χρειάζεται, αλλά δεν κολλάει πλέον με τον κανονισμό για τις προστασίες των δεδομένων. Και επιπλέον έχουμε έναν ορισμό που χρειάζεται για το e και τον χρειαζόμαστε πάλι το Electronic Communication Code και σχετίζεται πάλι με το ψηφιακό περιεχόμενο και τις υπηρεσίες μηνυμάτων. Αυτό είναι κάτι το οποίο δύσκολα συντονίζεται στο ευρωκοινοβουλευτικό επίπεδο και έχουν εντύπωση ότι τελικά αυτή τη στιγμή χανόμαστε κάπου για το ποιος κάνει τι, που, πώς και πότε. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε, νομίζω, ε, ειδικά όσον αφορά και τα θέματα μετανάστευσης ε, βάσεων δεδομένων κτλ. Γιατί έχω την αίσθηση ότι έχουμε τελικά μια ιδέα αντί να σκεφτούμε επί της αρχής ποια δεδομένα χρειαζόμαστε και πώς θα τα εφαρμόσουμε όλα αυτά για να ξέρουμε τελικά ποιος μπαίνει στην επικράτειά μας. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν ε, εμβαλωματικές ε, λύσεις. όπου βλέπουμε ότι δεν υπάρχει το θάρρος να κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει. Το ίδιο και στα ποινικά. Βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όπου λέμε επί της αρχής θα θέλαμε μια εισαγγελία που θα θα βοηθούσε την αστυνομία και το δικαστήριο, αλλά δεν καταλήγουμε ποτέ σε μια λογική να αποκτήσουμε ένα ποινικό σκέλος, τάξη ίσως να μην είναι και ρεαλιστικό. Αλλά αυτή η συνεχής ε, προσθήκη στοιχείων ε, οδηγεί σε ένα μοσαϊκό το οποίο δεν έχει συνοχή. Θα ήθελα λοιπόν λίγο περισσότερο θάρρος και εντάξει βεβαίως αυτό συνοφίλεται πιθανότατα και στο πολιτικό σκέλος αλλά χρειάζεται νομίζω θα έλεγα μια καλύτερη και πιο συνεκτική ενεολογική προσέγγιση των διαφόρων νομοθετημάτων. Thank you, Mrs. Ferrara. Η κυρία Ferrara. Grazie, Presidente. Grazie. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον Αντιπρόεδρο Τίμερμανς. Σήμερα μας μιλήσατε για μια ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση όπου πρέπει να βρούμε δραστικές λύσεις κατά του λαϊκισμού, της ξενοφοβίας, του εθνικισμού. 27 κράτη-μέλη γνωρίζουν τι θέλουν και θέλουν να προωθήσουν το κοινοτικό το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Εγώ συμμερίζομαι αυτήν την ε, δήλωση και θέλω να υπάρξει το ευρωπαϊκό εγχείρημα, το εγχείρημα της κοινότητας αυτής. Από τη στιγμή όμως που έφτασα στο Ευρωκοινοβούλιο πριν από τρία χρόνια, δύο θέματα συζητούνται διαρκώς και με αφήνουν πραγματικά ένα πορεία σε σχέση με την δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ακόμα δυστυχώς δεν την έχω δει. Πρώτα απ' όλα η προστασία που προκύπτει από την ε, Χάρτα των Θεμελιδών Δικαιωμάτων και δεύτερον, η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Σε ό,τι αφορά το πρώτο θέμα, θα θυμάστε ότι υπήρξε συγγήτρια για τη σχετική έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάσταση των θεμελιδών δικαιωμάτων 2014-2015. Και εκεί ήρθα αντιμέτωπη με κάτι που πραγματικά με άφησε άναβη Την ενεργοποίηση του άρθρου 7 σε περιπτώσεις παραβιάσεων συστηματικών περιστατικών που συμβαίνουν συχνά. Όταν ε, μιλάμε για θεμελιώδη δικαιώματα, πρέπει να δρούμε και προληπτικά, όχι απλώς να ερχόμαστε να θεραπεύσουμε καταστάσεις ε, που έχουν προκύψει ήδη και συστηματικά επαναλαμβάνονται. Σήμερα η ενεργοποίηση του άρθρου 7 δεν έχει λάβει χώρα ποτέ πήγε να γίνει λόγος όταν μιλούσαμε για την Ουγγαρία, αλλά δεν είναι σαφές πότε μπορεί να προληφθούν οι παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και για μένα αυτό είναι θεμελιώδου ε, σημασία. Η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων είναι αυτό που πραγματικά δίνει την νομιμοποίησή τη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ σα ρωτώ λοιπόν, τι πρόθεση έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προστατεύσει περισσότερο τα όσα προκύπτουν από τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, δηλαδή τα θεμελιώδη δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Και στην γνωμοδότηση της ε, επιτροπή ΛΥΜΠΕ, τη συναδέλφου Ιντβελτ για την παρακολούθηση, ε, με συγχωρείτε, αλλά δεν μας έχει πείσει πάρα πολύ η δημιουργία ενός μηχανισμού για την παρακολούθηση των χωρών που ενδεχομένως θα υπήρχαν απειλέ ή κίνδυνοι για την παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εγώ θέλω να καταλάβω επιτέλους πότε ενεργοποιείται αυτό το άρθρο 7 και τι συγκεκριμένα εργαλεία υπάρχουν για να προληφθούν οι παραβιάσεις των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Και για να έρθω στο δεύτερο σημείο, την ε, διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Και εδώ γίνεται λόγος ε, κάθε φορά για το ότι πρέπει να βρούμε λύσεις αποτελεσματικές. Οι λύσεις έχουν ακουστεί πολλές, έχουν απαριθμηθεί, υπάρχουν. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι στο να βρούμε τις λύσεις θεωρητικά, είναι στην βούληση που υπάρχει. Και εδώ αναφέρουμε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που σήμερα ουσιαστικά συγκεντρώνει τους εθνικούς εγωισμούς εγώ εργάστηκα για την τροποποίηση του κανονισμού του Δουβλίνου. Και έρχονται ειδήσει εντωμεταξύ ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θέλει να μπλοκάρει την αναθεώρηση του Δουβλίνου. Δεν θέλει καθόλου να προχωρήσει το θέμα, γιατί δεν υπάρχει στην ουσία συμφωνία για την κατανομή των ευθυνών. Στο πλαίσιο των διαθεσμικών λοιπόν σχέσεων και με σκοπό να βεβαιωθούμε ότι έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση ισχυρότερη. Εσείς τι θα μας πείτε σε σχέση με το Συμβούλιο και αυτή την έλλειψη πολιτική βούληση που υπάρχει. Πώ μπορούμε να ξεπεράσουμε την ε, έλλειψη πολιτική βούληση από την πλευρά των κράτων μελών. Ο πρόεδρο Γιούνκερ στην προηγούμενη Ολομέλεια έκανε λόγο για την ενεργοποίηση των επιπαραβάσει διαδικασιών που όμω δεν επιφέρουν ε, κυρώσει. Πώ να τερμινεύσουμε ότι δεν θα υπάρξουν καν κυρώσει. Ε, αυτό και μόνο το γεγονός ότι η συνεργασία θα είναι επιβεβλημένη δεν είναι ουσιαστικά απόδειξη αποτυχία του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Θα, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι αυτονόητο. Όχι να υπάρχει απειλή κύρωση. Θα θέλαμε λοιπόν να μα πείτε ποια είναι η δική σα άποψη και τι διαβλέπετε να συμβαίνει στο Συμβούλιο σχετικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για όλε. αυτές τι ερωτήσει Θα προσπαθήσω να απαντήσω στο καλύτερα μπορώ. Πολλοί ήταν οι λόγοι για την έκβαση που είχε το Βρετανικό Δημοψήφισμα. Να κάνουμε τώρα επιθανάτια αναφορά ε, και νεκροψία μπορούμε να το κάνουμε επί ώρες, αλλά αν επί 15-20 χρόνια λες ότι όλα τα κακά προέρχονται από τις Βρυξέλλες, που αφαιρούν το ένα, αφαιρούν το άλλο κτλ. Και μετά στο τέλος αυτής της κοτσαετίας ε, λες «Α, ξέρετε, παρεπιπτόντως, θέλουμε να ψηφίσετε υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Ε, δεν πρέπει να σας εκπλήσει τελικά που σας άκουσαν τις προηγούμενες δύο δεκαετίες ε, οι συμπολίτε σας. Το ενδιαφέρον που βλέπω να συμβαίνει τώρα είναι ότι ο κόσμος κατάλαβε ότι δεν, έχει, δεν είναι άμυρο επιπτώσεων ε, το να ε, θέλει κανείς να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή να κατηγορείς ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση συνέχεια και να λες ότι ό,τι είναι καλό είναι από την εθνική κυβέρνηση και ό,τι κακό είναι από τις Βρυξέλλες. Γιατί φάνηκε τώρα ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει και στο ενδεχόμενο αποτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση μακροπρόθεσμα. Κάποιοι αρχίζουν και λένε ότι ναι, μεν δεν μου ικανοποιούν όλα όσα γίνονται στι Βρυξέλλε, αλλά δεν θέλω και να ξεφορτωθώ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέτοια δείγματα βλέπουμε αρκετά. Νομίζω ότι αφυπνίζεται μια νέα πολιτική γενιά ε, στη, στον Άμενο Βασίλειο. Το είδαμε και στι τελευταίε εκλογέ. Πολλοί νέοι όμως ε, δεν σκέφτηκαν ε, όπως οι προηγούμενες γενιές. Το θέμα είναι τι ψήφισε ο καθένας. Αν οι νέοι δεν ψήφισαν, ε, δεν μπορούν και να παραπονούνται. Γιατί όποιο δεν ψηφίζει δεν μπορεί να παραπονείται εκ των υστέρων, για να μην πω κάτι άλλο. Είναι η στιγμή λοιπόν τώρα που όχι μόνο ίσως στην Ευρωπαϊκή Ένωση μάλλον στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γερμανία και αλλού βλέπετε οι νέοι να κατεβαίνουν στον δρόμο για να πούν ότι είναι σημαντικό για αυτούς το project αυτό, το ευρωπαϊκό Οικοδομήματο δηλαδή. Το σημαντικό είναι, θα σας πω τι πρέπει να γίνει. Δεν θέλω να πω κάτι για λαϊκισμό, γιατί δεν μου αρέσει αυτή η λέξη. Ας πούμε ότι έχουμε κάποιες αντιδραστικές ε, ή άκρο εθνικιστικέ δυνάμεις, οι οποίε συνδυάζουν δύο πράγματα. Επιθέτουν αυτό που λένε ότι είναι οι αξίε μα και το establishment. αντί να δημιουργηθεί ε, η εντύπωση ότι κάνουμε αυτό που θέλουμε, ότι δηλαδή προσπιζόμαστε τις αρχές μας, θεωρήθηκε ότι αγωνιζόμαστε για το establishment. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η ιδεολογική αντιπαράθεση. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Μην αυτά πατώμε. Θα έχουμε αφενός αυτούς που πιστεύουν στην ανοιχτή κοινωνία και αυτούς που πιστεύουν ε, στην κλειστή κοινωνία. Χάρη θρησκείας, ε, ιδεολογία ε, κτλ. κτλ. Ίσως το Brexit και η εκλογή του Τραμπ στις ΗΠΑ οδήγησε στην επίγνωση ότι η ψήφο έχει μία επίπτωση που μπορεί και να μην είναι η αναμενόμενη από τον ψηφοφόρο όταν έρχεται την ψήφο, όπως είδαμε με τις εκλογέ στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γαλλία, έτσι, να μην το ξεχνάμε και αυτό. Το ίδιο μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε. και υπάρχει κάποιο ο οποίο εκτίθεται κατά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνέχεια πρέπει να δούμε τι μέλλον θα έχει. Θα δούμε προ τα πού θα πάει το πράγμα. Για τι διαπραγματεύσει για το Brexit, δεν έχω να προσθέσω πολλά όσα έχουν υποθεί δημοσία. Για μας αυτό που είναι σημαντικό είναι να βάλουμε στην πρώτη γραμμή τα συμφέροντα των πολιτών μας και στο μυαλό μας και στην καρδιά μας. Δεν θέλουμε να υποφέρει κάποιος συμπολίτη μας και, δεν, και μιλώ και για τους Ευρωπαίους που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και για τους Βρετανούς που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερο σημείο που πιστεύω κράτονται πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Εγώ είμαι 56 ετών. Η συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής ήταν από, τα, από τους σταθμούς της δικής μου πολιτικής αντιδρομίας Πριν συμβεί κανείς δεν το πίστευε. Και κάτι που ποτέ δεν θα έπρεπε να συμβεί χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ευθύνη που ξεπερνά τις άμεσες ευθύνες. Είναι διαγενειακή ευθύνη, ώστε η συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής να παραμείνει μια επιτυχία. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, βλέποντας τα όσα συμβαίνουν. Στο νησί δίπλα στην Αγγλία δηλαδή και στη Βόρεια Ιρλανδία και στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Αυτό ξεπερνά τα άμεσα συμφέροντα. Δεν μιλάμε καν για τα φυσικά σύνορα, μιλάμε για μία από τις σημαντικότερες συνευτικές διαδικασίες τα τελευταία 40 χρόνια που ποτέ δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να απειληθεί από τις διαπραγματεύσεις ε, για το Brexit. Αυτό είναι το δεύτερο. Και το τρίτο, πιο γενικό, ευρύ σχόλιο, Ο Ιπποκράτης θα πρέπει να μας ε, καθοδηγεί. Ας κάνουμε το λιγότερο κακό, γιατί δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε κανέναν. Δεν το ζητήσαμε σε αυτό το διαζύγιο. Και προσωπικά εγώ εξέφρασα τη μεγάλη μου λύπη. Είναι τραγωδία. Αλλά συνέβη και έχουμε ευθύνη να μην προκαλέσουμε μεγαλύτερη ζημιά από την απολύτως αναγκαία σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. τώρα το Brexit δεν οδήγησε σε μια σειρά άλλων χωρών που εξέφρασαν το ίδιο αίτημα, δεν είχε αποτελεσμα ένα ντόμινο αποχωρήσεων. Θα πρέπει να δούμε και τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ διαφόρων κρατών, Ουγγαρία, Πολωνία. Αλλά δείτε και τι μεγάλη υποστήριξη, λαϊκή υποστήριξη υπάρχει στις χώρες αυτές για τη συμμετοχή στην Ένωση. 80% και παραπάνω. Μπορεί δηλαδή να διαφωνούμε σε κάποια πράγματα, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον. Όπως και η καμπάνια του Όρμπαν Stop Brussels, σταματήστε τις Βρυξέλλες. Αν δείτε το μετρό της Βουδαπέστης τώρα, που χρηματοδοτήθηκε και με κάποια κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά λέει, λέει ο Μπόρμπαν σταματήστε τις Βρυξέλλες. Είναι λίγο περίεργο όλα αυτά. Μετά όμω τι λέει μετά την καμπάνια του, Α, η Ουγγαρία είναι μια περήφανη ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί το λέει αυτό, γιατί ξέρει πολύ καλό ο κ. Σόρμπαν ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Ουγγρών γνωρίζουν ότι αξίζουν, ότι, συγγνώμη, ότι ανήκουν σε αυτή την ευρωπαϊκή οικογένεια. Άρα τα πράγματα δεν είναι άσπρο μαύρο. Υπάρχουν πολλέ απαντήσει σε αυτή τη συζήτηση και δεν νομίζω ότι στη Τσεχία έπαιξε και μεγάλη ανταπόκριση όταν ο Βάτσλαφ Κλάου είπε αυτά που είπε. Τι είχε πει, τσέξι, τσεκάου τέλο πάντων, όπω το πει. Τη μέρα μετά, αφού το είχε πει, μου στην Πράγα και δεν είδα να συγκινήθηκε και ιδιαίτερη κοινή γνώμη. Το ωραίο με την Τσεχία είναι ότι περισσότερο περισσότεροι Τσέχοι που γνωρίζω έχουν βαθιά ριζωμένη την αίσθηση της ηρωνίας, βλέποντας τον κόσμο και την πραγματικότητα. Και το ίδιο αυτό το αίσθημα το χρησιμοποιούν, όπως στην περίπτωση των παρατήρησεων του Βάτσλαβ Κλάους. Και βέβαια υπήρχαν κάποιοι που ήταν κατά. Πάντως υποστήριξη μετά το Brexit, ε, όπως έδειξε η ειδοσκόπηση στο Ευρωβαρόμετρο, έδειξε ότι αυξήθηκαν αυτοί που θέλουν την Ένωση και μετά τις εκλογές Τραμπ. Την εκλογή του Τραμπ. Για την ε, κοινότητα δικαίου, το κράτος δικαίου που είπε η κυρία Κάουφμαν. Όταν είπε ο κύριος Λεμπρετών Εσωτερικές υποθέσεις Πολωνίας. Τι σημαίνει μια οργάνωση που διέπεται από το κράτος δικαίου. Σημαίνει, όπως εμείς, υπογράφεις μια συνθήκη και την επικοινωνία και από εκεί και πέρα γίνεται δεσμευτική για σένα αυτή η συνθήκη. Δεν μπορείς απλά να πεις. Με βάση την εθνική κυριαρχία, ναι, υπάρχει αυτή η συνθήκη, αλλά ξέρετε, α, υπάρχει και εθνική Κυριαρχεί και εγώ διαλέγω ό,τι μ' αρέσει από τη συνθήκη και εφαρμόζω ό,τι θέλω εγώ με βάση την εθνική κυριαρχία. Η ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος είναι πολύ θεμελιώδη ζήτημα. Αν υπάρχουν αμφιβολίες για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, σημαίνει παραμέληση ε, χρέους, καθήκοντος εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην το ψάξει. Και νομίζω ότι η ανεκκρατησία της δικαιοσύνης μπορεί να πάρει πολλές μορφές. Αλλά σημαίνει ότι οι νομοθετικές εξουσίες και τελικές εξουσίες δεν ελέγχουν τα δικαστήρια. Αυτό νομίζω ότι είναι συμπεφωνημένο. Αυτή είναι η αρχή. Αν υπάρχουν στα κρατη με κινήσεις προς τη δημιουργία περισσότερου κρατικού έλεγχου πάνω στα δικαστήρια, πρέπει κάποιο να υψώσει τη φωνή του. Και αυτό το κάνω εγώ εδώ και 1,5 χρόνο με την υποβολή συστάσεων. Αλλά δεν έδειξε κάτι τέτοιο να οδηγεί σε μια προφανή αλλαγή πορεία τη κυβέρνηση. Είχαμε και ένα Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων πρόσφατα, όπου φάνηκε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών θα ήθελε η πολεμική κυβέρνηση να κάτσει στο τραπέζι με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη λύση του προβλήματος που έχει προκύψει. Και ελπίζω να πάρω κάποια μηνύματα από την πλευρά της Βαρσοβίας, ώστε να μας δείξουν ότι θέλουν και αυτοί να αποφύγουν περαιτέρω συστηματικές απειλές ε, στο κράτος δικαίου. Κάτι που δυστυχώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Αν αυτό τώρα σημαίνει παρέμβαση στα εσωτερικά της Πολωνίας, όταν υπάρχει ζήτημα ανταγωνισμού, και πρέπει να ληφθούν μέτρα από εμάς. Γιατί αυτό κάνουμε εμείς ως Επιτροπή. Όταν υπάρχει θέμα κρατικών ενισχύσεων πρέπει να παρέμβουμε. Αυτή την εντολή μας την δίνει η συνθήκη. Την έχουν γράψει και επικυρώσει όλες οι χώρες μέλη αυτή τη συνθήκη. Στην περίπτωση της Ουγγαρίας. Γιατί και για την Ουγγαρία, κύριε Λεμπρετών, κάνατε μια ερώτηση. Υπάρχει διαδικασία επί παραβάση. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει ως Κομισιόν τη θέση μας η Ουγγρική κυβέρνηση θα έχει κάθε ευκαιρία να μας πει την άποψή της και θα δούμε πού αυτό θα μας οδηγήσει. Σε κάθε διαδικασία, γιατί υπάρχουν πολλές μετακρατημέλη, αυτό συμβαίνει. Την προηγούμενη εβδομάδα δρομολογήθηκε μια διαδικασία προς την Ουγγαρία, αλλά και μια χώρα που ξέρω πολύ καλά, την Ολλανδία. Άρα Υπάρχουν διαδικασίε επί τακτά διαστήματα, κατά κρατομήλων. Αυτό είναι ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και από τη στιγμή που έχει κινηθεί αυτή η διαδικασία, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να επισέλθω σε λεπτομέρειες πάνω στην περίπτωση που αναφέρατε, γιατί τώρα έχει ξεκινήσει ο διάλογος με την Ουγγρική κυβέρνηση. Το ίδιο με τον νόμο για το άσυλο. Στείλαμε μια επιστολή ε, προειδοποίησης στις Ουκρικές Αρχές και για αυτό το θέμα. Τώρα επανέρχομαι στην επιτροπολογία. Εγώ θα ήθελα να έχουμε σημειώσει περισσότερη πρόοδο στο θέμα αυτό, αλλά επειδή έχω ασχοληθεί με το θέμα αυτό εδώ και 20 χρόνια, διάφορες μορφές του, γνωρίζω πως πάντα θα υπάρχει μια διελκυστίνδα μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου, γιατί ο ΜΕΝ προτιμά πράξεις ε, κατά εξοδότηση, η προτιμούν ε, πράξεις εφαρμοστικές, η Κομισιόν προτιμάει μια ε, λύση η οποία θα λειτουργεί και όχι να αποφασίζουμε εμείς όταν δεν μπορούν να αποφασίσουν τα κράτη-μέλη. Όλοι ξέρετε το θέμα των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, του, της γλυφωσάτης δεν μπορούν να συμφωνήσουν και τα πασάρουν στην Κομισιόν. Όχι επειδή θεωρώ ότι είναι κακό για την Κομισιόν, είναι κακό, αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος. Ο λόγος είναι ότι δημιουργείται έτσι η εντύπωση στη δημόσια γνώμη πως υπάρχει κάτι το οποίο εμείς δεν θέμε, αλλά οι Κομισιόν και οι γραφειοκράτες των Βρυξελών μας το επιβάλλουν. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι τον Ζαν Κλοντιούν και να λέει φτάνει πια. Δεν θέλω αν θέλετε η γλυφοσάτη να παραμείνει με βάση τα επιστημονικά στοιχεία, βγείτε και πείτε το. Και μην λέτε, α, δεν φταίω εγώ, φταίει η Κομισιόν ε, και τα λοιπά. Έχουμε δύο στόχους λοιπόν. Πρώτον, να προσπαθήσουμε να βρούμε έναν συμβιβασμό μεταξύ Κοινοβουλίου και ε, Συμβουλίου και βεβαίως ε, δεύτερον να δημιουργήσουμε ένα σύστημα στο οποίο ο κόσμος θα αναλαμβάνει την ευθύνη για τις θέσεις του και δεν θα απεκδίεται αυτή της ευθύνης. Για τους ε, καταγγέλλοντες. Ε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πάνω σε αυτό δουλεύουμε. Ξέρετε ότι ολοκληρώθηκε πρόσφατα η διαβούλευση, για εδώ, το λένε και τα χαρτιά μου. Ε, λάβαμε 6.000 απαντήσεις. 200 από διάφορες οργανώσεις. Οπότε υπήρχαν και πολλές άμεσες απαντήσεις, όχι μόνο από τις οργανώσεις, άρα οι περισσότερες από τους πολίτες. Το αναλύουμε και ακούμε πολύ προσεκτικά τις συζητήσεις. Οπότε πείτε μας κι εσείς τι θέλετε να κάνουμε. Να μας ε, βοηθήσει να καθορίσουμε και την πρόταση. Και άκουσα πολύ προσεκτικά τις ε, παρατηρήσεις που έγιναν. το θέμα του κυρίου Άντερσον ε, για το τι θα γίνει αν αλλάξει γνώμη το Ηνωμένο Βασίλειο. Κοιτάξτε, ε, δεδομένων των συνθήκων που επικρατούν, ε, πιθανότερο είναι να βγει ο ήλιος από τη Δύση παρά να αλλάξει θέση το Ηνωμένο Βασίλειο. Το τι είπε ο κύριος Φερχόφστατ είναι θέση του κύριου Φερχόφστατ, έτσι. Και είναι τελείως υποθετικά πράγματα. Εγώ προσωπικά θα δεχόμουν το Ηνωμένο Βασίλειο με ανοιχτές αγκάλες αν αποφάσιζε να ξανάρθει. Αλλά δεν το βλέπω, ειλικρινά. Είχαμε κάποια ξεκάθαρα μηνύματα πάλι από τον κύριο Ντέιβις σήμερα. Θα συμβεί. Όσοι παρακολουθούμε το Ηνωμένο Βασίλειο στενά, το ξέρουμε ότι θα συμβεί. Το θέμα είναι το πώς θα γίνει και τι ακριβώς θα συμβεί. Ελπίζω να έχουμε κάποια ε, σαφήνεια από την κυβέρνηση της αυτής μεγαλειότητας προσεχώς. Αλλά αυτό είναι μια υπόθεση εργασίας. Αυτή είναι η υπόθεση εργασίας ε, για την Κομισιόν. Λοιπόν. Συνοχή, είπατε, τις νομικές δράσεις. Κύριε Φως, συμφωνώ μαζί σας. Ε, το πρόβλημα είναι δυσυπόστατο. Το ένα είναι ότι εργαζόμαστε επί τη βάση 27-28 συγκρίσιμων μεν, αλλά διαφορετικών νομικών συστημάτων με προϋπάρχουσα συχνά νομοθεσία. Λοιπόν, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Καλό θα ήταν να υπάρχει τάμπουλα ράζα, αλλά δεν γίνεται. Υπάρχει πολιτική πραγματικότητα. Και όπως ξέρετε, σε όλους αυτούς τους τομείς ε, μπαίνουμε σε μια διαπραγμάτευση. Όλοι ξεκινάνε με διαφορετικές θέσεις και τελικά θα πρέπει να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση και νομίζω ότι και οι δυο μας ε, θέλουμε ο συμβιβασμός να λειτουργεί τελικά για τον πελάτη, για τον τελικό καταναλωτή. Και εκεί πέρα έχω τις ανησυχίες ε, μου, γιατί συχνά λόγω των διαπραγματεύσεων το γεγονός ότι υπάρχει συμβιβασμός είναι πιο σημαντικό από το ότι, ε, από το περιεχόμενό του. Και τελικά αυτοί που την πληρώνουν αυτοί που πρέπει να εργαστούν με αυτή την ομοθεσία. Οι καταναλωτές, αν θέλετε, οι πολίτες δηλαδή, οι, οι εταιρείε, ε, οι αρχέ Γι' αυτό και προέκυψε και η πρότασή μας ε, για την καλύτερη νομοθεσία. Γι' αυτό ζητήσαμε ακριβώς μια αξιολόγηση αντικτύπου, όχι μόνο για την πρόταση Κομισιόν, αλλά και για το αποτέλεσμα του συμβιβασμού. Γιατί η μόνη πρόταση που έχουμε τώρα είναι η λεγόμενη πυρηνική λύση. Να αποσύρουμε την πρόταση αν θεωρούμε ότι το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων έχει απομακρυνθεί πολύ από τον αρχικό φορέα. θα ήθελα κάποιο εξωτερικό ανεξάρτητο να πει όταν έχουμε ένα συμβασμό, εάν αυτό είναι ακόμα λειτουργικό και εφαρμόσιμο. Για τα συγκεκριμένα ζητήματα που θέσατε, ηλεκτρονική ιδιωτικότητα κτλ. Θα δείτε τον συνάδελφο τον κύριο Άντσιπ, δεν θα έρθει. Ναι, αυτός τα ξέρει καλύτερα αυτά. Τα ζητήματα, τα συγκεκριμένα. Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ... Α, ναι, ναι, η ώρα περνάει. Στο θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ήδη αναφέραμε κάποια από αυτά στο άρθρο Να πω κάτι ακόμα. Αυτό λειτουργεί μόνο εάν όλοι αισθάνονται ευθύνη. τα τελευταία χρόνια σε πολλές περιπτώσεις ε, θα με είχε πρωτοσέλιδο όχι μόνο η Γκαζέτα Βιμπόρζα αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα με είχαν αποθεώσει εάν είχα ξεκινήσει το άρθρο 7. Δεν θα άλλαζε τίποτα γιατί δεν θα είχαμε στήριξη στο Συμβούλιο για να κάνουμε κάτι αλλά αυτή είναι μια πολιτική πραγματικότητα την οποία πρέπει να αντιμετωπίσω. Εξακολουθώ να θεωρώ ακόμα και μετά από όλε τις προσωπικές επιθέσεις που δέχομαι κάθε μέρα θεωρώ ότι ο διάλογος είναι ο καλύτερος τρόπος για να λύσουμε αυτό το ζήτημα. Αλλά ο διάλογος θα λειτουργήσει μόνο εάν τα κράτη-μέλη αντιληφθούν ότι και τα, και τα άλλα κράτη-μέλη πρέπει να θέλουν να λειτουργήσει κάτι και να στηρίξουν την Κομισιόν για να μπορέσουμε έτσι να βρούμε μια λύση. Και εκεί καμιά φορά, το θέμα ότι το κάθε κράτος μέλος ζει ε, σε γυάλινο πύργο. Ε, δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, θα πρέπει να έχουμε το θάρρος όταν κάτι δεν λειτουργεί να το πούμε. Γιατί ασχολούμαστε τόσο πολύ και είμαστε πολύ καλοί στο να βρίσκουμε τα προβλήματα υποψηφίων χωρών, αλλά όταν ε, μπούμε μέσα είναι λίγο δύσκολο να μιλήσουμε για αυτά τα ζητήματα. Είναι και θέμα βεβαίως του Χάιντερ ε, και το ότι δεν μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε το FPE και την κυβέρνηση της Αυστρίας. Ε, εξακολουθεί να υφίσταται. Οπότε θα πρέπει τα κράτη-μέλη όλα να δουν ε, το ζήτημα με ένα πνεύμα συνεργασίας. Ελπίζω λοιπόν να μας βοηθήσει αυτό και επίσης θεωρώ και το είδα αυτό και στην κυρία Ινετφέλτ η οποία δεν ζήτησε νέες δομές, αλλά είπε ότι πρέπει να συντονιστούμε καλύτερα. Εδώ. Είμαι ο άνθρωπός σας λοιπόν. Αν αυτό θέλετε, είμαι στην διάθεσή σας για το πώς θα συντονίσουμε καλύτερα τα υφιστάμενα. Δηλαδή, το να κοιτάμε την εφαρμογή του κράτου δικαίου είναι κάτι το οποίο κάνουμε για όλα τα κράτη-μέλη. Υπάρχει μια ίση αντιμετώπιση για το θέμα της μετανάστευσης. Χρειάζεται συνένεση μεταξύ των κρατών μελών, αλλά μιλάμε, ε, είναι κάτι το οποίο αφορά την καρδιά των κρατών μελών και το ξέρουμε αυτό και αποδίδει πολιτικά να ασχολείται κανείς με τους φόβους των ανθρώπων την τρομοκρατία, η τρομοκρατία συνδέεται με τη μετανάστευση και ειδού ε, αυτή την κατάσταση αντιμετωπίζουμε Ελπίζω λοιπόν να συνεργαστούμε και να βρεθεί μια διέξοδος. Ε, το θέμα των ποσοστώσεων είναι ένα μικρό κομμάτι του Μπάζλ σε μια πολύ εξαιρετική κατάσταση κρίσεως. Τα πραγματικά πράγματα που χρειάζεται να κάνουμε είναι η προστασία των εξωτερικών σύνορων, καλύτερες συμφωνίες με τις χώρες στην Αφρική και καλύτερη πολιτική επιστροφής, ένταξης ε, στις χώρες μας και μετά, αν για κάποιον λόγο ένα ή δύο κράτη-μέλη, όπως είναι το 2015 με την Ελλάδα και την Ιταλία, πλημμυρίσουν από μια τεράστια διεθνή κρίση, να μην εφαρμόσουμε τον παραδοσιακό κανονισμό του Δουβλίνου για να τους πούμε «Α, δικό σας πρόβλημα». Αλλά πρόκειται για πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις. Ε, δεν αντιλαμβάνομαι. Έχω πρόβλημα μετά να λένε ε, μετά κάποιοι ηγέτες να λένε οι Βρυξέλλες μας επιβάλλουν να αλλάξουμε τον πολιτισμό μας γιατί θα πάρουμε μερικές χιλιάδες άτομα που θα τα επιλέξουμε εμείς. Πρέπει να είμαστε κάπως πιο ειλικρινείς. Γιατί μπορεί να γίνει αυτό. Ας το δούμε και την άλλη πλευρά. Χώρες όπως η δικιά μου. Που έχουν ε, εμπειρία στο θέμα ετών δεν είχαν αρκετή επιτυχία στο θέμα της ένταξης. Και το γεγονός ότι κάποιοι τώρα θεωρούν ότι μπορούν να σκοτώνουν τους συμπολίτε τους ε, ε, τζιχαντιστικά ε, είναι άτομα δεύτερης τρίτης γενιάς από τη Γαλλία, τη Βρετανία κτλ. Και ένα πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και άλλες χώρες λένε εφόσον δεν το έχετε καταφέρει εσείς ανησυχώ και εγώ, αυτό το αντιλαμβάνομαι. Αλλά από εκεί να πούμε δεν θα πάρω λίγες χιλιάδες γυναικόπαιδα, ε, αυτό με ξεπερνά. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ελπίζω να μπορέσει να, να κάνουμε μια συζήτηση επί του θέματος, ειδικά με τις ε, χώρες αυτές ε, που είναι τόσο κάθετες για το θέμα αυτό. Με συγχωρείτε που ακρηγόρησα. Το παράκανα, ελπίζω να μην σας πείραξε. Ευχαριστώ λοιπόν. Uh, uh, uh, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε πρώτα αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κύριε Τίμερμανς. Η συζήτηση που είχαμε ήταν στο πλαίσιο του διαθεσμικού διαλόγου που έχουμε. Προσβλέπω και στην επόμενη συνάντηση. Γιατί Λίγοι μεν ήμασταν ε, στην αίθουσα, αλλά παρόλα αυτά υπήρξε μια πολύ πλούσια ανταλλαγή απόψεων. Σας ευχαριστώ για αυτό λοιπόν. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε μέρα μας. colleagues, continue by item number and I would like to give the floor. Ευχαριστούμε. Να περνάμε στο επόμενο σημείο τη Περιφερειακή Διάταξη. Θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο τη Νομική Υπηρεσία για να μα παρουσιάσει το διοργανικό εγχειρίδιο για την σύνταξη νομοθετικών πράξεων. Παρακαλώ να είστε σύντομο όμω, γιατί 15 λεπτά πίσω είμαστε ήδη στο χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ιδίω δε που μου τον δίνετε αμέσως μετά την επίσκεψη του κυρίου Τίμερμανς που μας μίλησε για την καλύτερη νομοθεσία που ανήκει στο χαρτοφυλάκιό του. Εγώ είμαι εδώ για να σας παρουσιάσω αυτό τη νέα δημοσίευση για το διοργανικό εγχειρίδιο τη νομοθετικών πράξεων στο πλαίσιο τη κανονική ε, νομοθετική διαδικασία. Ο τίτλο είναι μακρύ και μα λέει όμω ε, ότι αυτή, αυτό το εγχείρημα έχει και τα ωριά του, αλλά είναι και φιλόδοξο. Είναι ένα εγχειρίδιο. Άρα πρέπει να είναι εύκολο, να μπορεί κανείς να το συμβουλεύεται γρήγορα. Είναι ένα κοινό για τα τρία θεσμικά όργανα, Συμβούλιο, Κομισιόν ε, και Κοινοβούλιο. Αντικαθιστά τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή τα εσωτερικά έγγραφα που κάποιε φορέ αποκλίνουν μεταξύ του και που αποτελούν μοντέλο γιατί, που, έχουν, που είναι υποδείγματα σε κάθε κράτος, ε, σε κάθε θεσμικό όργανο. Πρόκειται για τη μορφή των ε, νομοθετικών πράξεων, αλλά χωρί τη μορφή, χωρί τον τύπο δεν μπορούμε να έχουμε και περιεχόμενο. Η παρουσίαση δεν θέλουμε να τα ρυθμίσουμε όλα. Ακολουθούμε το τι προβλέπεται για την τακτική διαδικασία. Άρα, ό,τι αφορά την τακτική νομοθετική διαδικασία περιλαμβάνεται σε αυτό το χείρι, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα, αλλά περιλαμβάνονται οι βασικέ δραστηριότητε νομοθετικέ στο πεδίο εφαρμογή. Το εγχειρίδιο είναι αποτέλεσμα εργασία ενό τεχνικού οργάνου, ομάδα διοργανικού προβληματισμού νομοθετικού, νομοτεχνικού περιεχομένου. Σε ό,τι αφορά το Κοινοβούλιο, περιλαμβάνονται εκπρόσωποι της νομικής υπηρεσίας και, τη γάμα δέλτα Προεδρία για το, την του Κοινοβουλίου. Όποιοι ξέρουν τον κοινό πρακτικό οδηγό για όσους συνεισφέρουν στις εξωματικών πράξεων, τον Γκρίτλ, από την τελευταία έκδοση του 2013 έχει αναλάβει η ομάδα να αλλάζει αυτό το κοινό εγχειρίδιο. Ήδη το έχει αλλάξει. Το γκρίτλ αυτό το εγχειρίδιο. Με κάποιες ε, εκφράσεις οποίες μπορούν να χρησιμοποιούνται το πλαίσιο κάποιων ε, νομοθετικών πράξεων που θα τους οπισθακτήσεις της νομοθετική διαδικασία έχουμε για τη γαλλική και αγγλική εκδοχή και τις μεταφράσεις. Ελέγξαμε ενδελεχώς τις μεταφράσεις. Τέσσερα πλαίσια το εγχειρίδιο, έχει και ένα παράρτημα. Το πρώτο τμήμα είναι ένα υπόδειγμα νομοθετικής πράξης, το δεύτερο είναι νομοθετική εξέταση που είναι ένα τυπικό, τυπική μορφή, ένα τυπικό υπόδειγμα. Υπάρχουν επίσης κάποια τα κανόνες διατύπωσης. Εκεί μιλάμε για την ανάθεση εκτελεστικών και άλλων αρμοδιοτήτων, ορισμούς, τροποποίηση πράξεων, ε, έναρξη ισχύω, εφαρμογή και δικαιούχους. Αυτά τα υποδείγματα δεν τα έχουν φανταστεί τα μέλη του Γκρίτλ, αλλά τα έχουν συλλέξει από διάφορα έντυπα, όπως η Συμφωνία για την Νομοθεσία του 16 ή μια άλλη συμφωνία για την ποιότητα της διατύπωσης του 98. Και φυσικά λαμβάνουν υπόψη τις συνθήκες και την ομολογία. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι αλλάζει το καθεστώς ε, του εγχειριδίου ή, αυτής της, ε, ή αυτού του υποδείγματος εντύπου. Απλά είναι εύκολο να τα εντοπίζουμε με συστηματικό τρόπο τα διάφορα αυτά υποδείγματα. Και βέβαια κυρίως χρησιμοποιείται ηλεκτρονικά αυτό το εγχειρίδιο και περιλαμβάνει υπερσυνδέσεις ε, hyperlinks. Κάθε μέρα αναεπικαιροποιείται. Άρα είναι μια εργαλειοθήκη. Φυσικά τα θεσμικά όργανα, αν θέλουν ε, ή κρίνουν ότι η κατάσταση το απαιτεί, μπορούν να μην χρησιμοποιήσουν αυτά τα υποδείγματα. οι μεταφραστικές υπηρεσίες θα βρουν όλες τις ε, εκφράσεις σε διάφορα τεχνικά λεπτά ζητήματα για θέματα που επαναλαμβάνονται, που επανέρχονται. Σίγουρα θα υπάρξει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου από αυτό το νέο εγχειρίδιο. Ευχαριστώ. Ε, thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουν οι συνάδελφοι τίποτα σχόλια για την παρουσίαση. Δεν φαίνεται να έχετε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας και περνάμε στο σημείο 6. Ανταλλαγή απόψεων για την ηλεκτρική δημοσίευση της εφημερίδας των Ευρωπαϊκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την οποία είμαι εισηγητή, πολύ γρήγορα να συνοψίσω το τι συμβαίνει. Μιλούμε για μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στόχο έχει να θεωρήσει τον κανονισμό 2.16 κάθετος 2013 για την ηλεκτρονική δημοσίευση της επίσημης εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ε, καθορίζει τον κανόνα ότι η ηλεκτρονική δημοσίευση ισοδυναμεί με την εξορισμού έγκυρη έκδοση της επίσημης εφημερίδας και ότι η έντυπη δημοσίευση της επίσημης εφημερίδας θα έχει νομική ε, νομικό κύρος ή αξία σε έκτακτες ε, συνθήκες και την προσωρινή περίπτωση διακοπής της ηλεκτρονικής δημοσίευσης. Η αλλαγή αυτή σκοπό είχε να ε, ενισχύσει την νομική βεβαιότητα βελτιώνοντας την πρόσβαση στην επίσημη εφημερίδα και για να μπορούν όλοι να δίνουν πίστη στην ηλεκτρονική εκδοχή της εφημερίδας και όχι στην έντυπη ε, έκδοσή της. Ο κανονισμός επιπλέον προβλέπει η ηλεκτρονική δημοσίευση της επίσημης εφημερίδας να έχει μία προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή βάσει της οδηγίας 1999 κάθετος 93 κάθετος ΕΚ σε ένα κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές. Η οδηγία αυτή έκτοτε έχει ε, ακυρωθεί και αντικατασταθεί από τον κανονισμό υπαριθμών 9-10 κάθετος 2014 που εισάγεται δυνατότητα επίσημης έγκρισης εγγράφου με μία προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα βάσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το άρθρο 353 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αποκαλούμενη ρήτρα ευελιξίας, η οποία χρησιμοποιήθηκε για τον κανονισμό που πρόκειται να τροποποιηθεί, είναι αυτή που επιτρέπει να υπάρξει διαδικασία της συγκατάθεσης, όπου το Κοινοβούλιο έχει στη διάθεσή του δύο επιλογές. Μπορεί είτε να εγκρίνει είτε να απορρίψει την πρόταση. Η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, εφόσον δει, μπορεί να υποβάλει και σχετική έκθεση, συμπεριλαμβάνοντας ένα ψήφισμα μη νομοθετικού χαρακτήρα, απαριθμώντας τους λόγους, την αιτιολόγηση δηλαδή που το κοινοβούλιο μπορεί να προσφέρει ή να αρνηθεί τη συγκατάθεσή του, προβλέποντας συστάσεις για την υλοποίηση της προτινόμενης πράξης. Η προτινόμενη τροπολογία βεβαίως έχει βασιστεί σε νέες διατάξεις για τις ηλεκτρονικές σφραγίδες βάσει του ανοθη αναφερθεντος αναφερθέντος κανονισμού υπαριθμών 910-2014, ο οποίος εγκρίθηκε βάσει της τακτικής νομοθετικής διαδικασίας, δηλαδή συναπόφαση, βάσει του άρθρου 114 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εναρμόνιση μέτρων στην εσωτερική αγορά. Αυτό εγείρει το ερώτημα για το κατά πόσον νομική βάση για την αναθεώρηση του κανονισμού 216 κάθετος 2013 για την ηλεκτρονική δημοσίευση της επίσημης εφημερίδας θα έπρεπε να είναι η ρήτρα ευελιξίας. Αυτά είναι τα στοιχεία και το θέμα που μας απασχολεί. Έχετε καθόλου σχόλια συνάδελφοι. Κυρία Κάφμαν, θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω ένα ερώτημα, γιατί δεν είμαι σίγουρη, εάν κατάλαβα καλά. Ε, ως εισηγητής, ήσασταν υπέρ, ε, ή τι είπατε τώρα, υπέρ μιας ε, έκθεσης πρωτοβουλίας. Ή είπατε μόνο ότι υπάρχει δυνατότητα να γίνει κάτι τέτοιο. Ήταν α, κάποιες αρχικές σκέψεις, εάν θέλετε. Και θα υπάρξει ένα σχέδιο έκθεσης και θα επανέλθουμε μετά σε αυτό. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Σεβέρ από την υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ένωσης και ο κύριος Γκρίγκολόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλετε τον λόγο. Ευχαριστώ, Εμμανουέλη Γκριγκολόν. Σύντομα, έξω όσων ξέρουμε και από τις ε, πληροφορίες που λάβαμε από συναδέλφους στο Συμβούλιο, σκοπεύουν ε, να το δουν αυτό στο δεύτερο μέρος της Προεδρίας ε, της Εστονίας. Αυτά για όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχουν σχόλια ε, με την συμφωνία της Επιτροπής ε, προτείνω να επαληθεύσουμε την νομική βάση της πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 39 του κανονισμού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ συνεχίζουμε με το σημείο υπαριθμών 7. Εξέταση σχεδίου έκθεσης ε, για την εφαρμογή της οδηγίας 2004 35 κάθετος ΕΟΚ. Τον λόγο έχει η κυρία Φεράρα που είναι η συγγήτρια. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μετά από έξι μήνες εντατικής εργασίας επιτέλους φτάσαμε στην παρουσίαση της ε, πρότασης ε, για την έκθεση για την περιβαλλοντική αστική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την διόρθωση της ζημιάς στο περιβάλλον. Στόχος είναι να υπάρξει μια κοινή ευθύνη, όπως είπαμε, για τα ζητήματα αυτά. Βασίζεται στην αρχή ο Ριπένον πληρώνει του άρθρου 191 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η οδηγία περιέχει έναν γενικό ορισμό της περιβαλλοντικής ζημίας, δηλαδή μετρήσιμη μείωση της ποιότητας μια, ενός φυσικού πόρου ή της δυνατότητας χρήσης του που μπορεί να έχει άμεσα ή έμεσα αποτελέσματα και υπάρχει και άλλη μία κατηγορία ζημίας ε, που αφορά την βλάβη σε απειλούμενα είδη, τη βλάβη στα ύδατα και στο έδαφος. Ε, έχουμε εδώ πέρα λοιπόν διάφορες πηγές οποίες βασιστήκαμε, εκθέσεις της Κομισιόν, ειδικών, αλλά επίσης και τις παρεμβάσεις των ειδικών που συλλέξαμε κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου που οργανώσαμε με τον ε, κύριο Γιάβορα από την Γενική Διεύνηση Ένβη της Κομισιόν η οδηγία λοιπόν εφαρμόζεται σε όλες τις εταιρείες οι οποίες κατά διάρκεια των δραστηριοτήτων τους προκαλούν ή θα μπορούσαν να προκαλέσουν ε, βλάβη στο περιβάλλον. Πέρα από αυτές τις ε, δραστηριότητες ε, πρέπει να δούμε και να εξετάσουμε και την συμπεριφορά η οποία είναι βλαπτική προς το περιβάλλον κατά την άσκηση κάποιας ε, επαγγελματικής δραστηριότητας. Οπότε πρόκειται για πολύ περιορισμένο πεδίο εφαρμογής, δηλαδή αφορά συγκεκριμένο τύπο ε, βλάβης προς το περιβάλλον, έδαφος, νερό και βιοπικιλότητα και μόνο για συγκεκριμένες δραστηριότητες οι οποίες ε, θεωρούνται επικίνδυνες και περιέχονται σε έναν συγκεκριμένο κατάλογο. Υπάρχει λοιπόν, θα έλεγα, μία αβεβαιότητα όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή της ε, οδηγίας, ειδικά στο θέμα της ευθύνης που περιέχεται στο άρθρο 4. Έχουμε λοιπόν μια ανάλυση η οποία έχει γίνει σε διάφορες μελέτες της ε, Κομισιόν, ειδικά στο άρθρο 18 παράγραφος 2L. Ε, Έχουμε λοιπόν ένα κατακαιρματισμό και συχνά βλέπουμε ότι οι διατάξεις αυτές αποδεικνύονται αναποτελεσματικές. Τα βασικότερα κενά αφορούν την έλλειψη μιας συγκεκριμένης διοικητικής διοδικασίας ε, την οποία θα έπρεπε να υιοθετήσουν τα κράτη για να μπορέσουν ακριβώς να δουν αν υπάρχει ανάγκη να παρέμουν σύμφωνα με την οδηγία σε περιπτώσεις βλάβης ε, του περιβάλλοντος. Οπότε η μελέτη της Κομισιόν έδειξε ότι πολλά κράτη-μέλη, ακριβώς επειδή υπάρχει δυσκολία εφαρμογής ε, της σχετικής οδηγίας, χρησιμοποιούν το εσωτερικό τους δίκαιο για να αντιμετωπίσουν ε, τα ζητήματα αυτά ε, ζημίας στο περιβάλλον. Έχουμε λοιπόν έτσι ένα πεδίο το οποίο είναι αντιφατικό και μη ολοκληρωμένο και υπάρχει συγκεκριμένη δυσκολία για να έχουμε ένα εναρμονισμένο καθεστώς ε, οικονομικής εγγύησης. Και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι η οδηγία δεν έχει καθόλου κάποιες ε, προβλέψεις για το τι θα γίνει στην περίπτωση παραδείγματο χάρη που ο υπεύθυνο ή η έχει χρεοκοπήσει ή δεν μπορούμε να κρίνουμε ποιος είναι υπεύθυνο ε, για μια ζημία. Και το βάρος πέφτει τελικά στη δημόσια διοίκηση, δηλαδή στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, η οδηγία δεν αποκλείει τη δυνατότητα τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν αυστηρότερες ε, διατάξεις. Καλό θα ήταν λοιπόν να υπάρξει μια διάταξη που θα δημιουργήσει μια δευτερογενή ευθύνη σύμφωνα με τα υποδείγματα που υπάρχουν σε κάποια κράτη-μέλη, στην ε, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία κλπ. Παραδείγματο χάρη, εάν ε, κλείσει μια τέτοια εταιρεία και δεν είναι δυνατόν να βρούμε τον ε, υπεύθυνο, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις και αν υπάρχει κάποια διάδοχη μορφή. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από την οδηγία και θα μπορούσαν να καλυφθούν από τις συνήθεις εγγυήσεις όπως οι μεγάλες καταστροφές. Στην περίπτωση αυτή θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κάποια ευρωπαϊκά κονδύλια και οι νέες δυνατότητες που υπάρχουν στο τεχνολογικό και ιατρικό πεδίο μας δίνουν πώς υπάρχουν και επιδράσεις των βιομηχανικών δραστηριοτήτων στον ανθρώπινο οργανισμό. Υπάρχει έτσι κίνδυνος ε, της βιολογικής ισορροπίας ε, σε μεγάλο βαθμό περιπλοκότητας ε, και υπάρχει έτσι μια σειρά παραγόντων που μπορούν να παρέμβουν στον ανθρώπινο οργανισμό με πολύ καταστροφικό τρόπο. Για όλους αυτούς τους λόγους θα πρέπει ο νομοθέτης να προβλέψει την δυνατότητα αναδιατύπωσης της βλάβης προς το περιβάλλον, η οποία θα είναι ομοιογενής, αλλά και θα μπορεί να προσαρμοστεί στις διάφορες βιομηχανικές δραστηριότητες και τις βλάβες που προκαλούν. Και να υπάρχει η δυνατότητα να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογή τη οδηγίας και στη βλάβη στον αέρα, στην χλωρίδα και την πανίδα, στο τοπίο και να προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε τις νέες αυτές επικίνδυνες δραστηριότητες θα μπορούσαν να μπουν στον κατάλογο δραστηριοτήτων που ε, περιέχεται στην οδηγία. Σύμφωνα με τις έρευνες της ε, Κομισιόν και τις μαρτυρίες διαφόρων ενδιαφερομένων, προέκυψε πως ε, ήδη στις περισσότερες από τις περιπτώσεις η βιομηχανία έχει προβλέψει ένα σύστημα οικονομικών εγγυήσεων για τα όσα καλύπτει η οδηγία ELD και αυτό, σε αυτό συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας. Οπότε μπορούμε να βελτιώσουμε το πεδίο εφαρμογής ε, και έτσι θα γίνει πιο ξεκάθαρο το νομικό πλαίσιο και το πεδίο εφαρμογής οδηγίας. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα πράγματα θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιες διατάξεις οι οποίες ε, θα διευκολύνουν την ύπαρξη μιας διασφάλισης ε, για τις ε, περιπτώσεις αυτές, βασιζόμενη σε πολλές μελέτες ε, σκοπιμότητας που αφορούν ακριβώς τον υποχρεωτικό χαρακτήρα ασφάλισης έναντι τέτοιων κινδύνων των βιομηχανιών. Επίσης, θα μπορούσαμε να δούμε κάποια άλλα στοιχεία για να βελτιώσουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν εδώ πέρα. Να υπάρξει παραδείγματος χάρη ένα ευρωπαϊκό μήτρο για τις περιπτώσεις ELD και για τις εταιρείες οι οποίες ασκούν επικίνδυνες δραστηριότητες. Βάσει του παρατήματος 3 της οδηγίας με τη θέσπιση ενός συστήματος οικονομικού ελέγχου για τους φορείς που έχουν επικίνδυνες ε, δραστηριότητες. Επίση, οι φραγμοί στην υλοποίηση τη οδηγία έχουν να κάνουν με την ελληπή προετοιμασία των εθνικών αρχών, που δεν είναι πάντοτε σε θέση να υλοποιήσουν αποτελεσματικέ διαδικασίε για να αντιμετωπίσουν του υπευθύνου των περιβαλλοντικών ζημιών. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να σχεδιάσει και να στοχεύσει το πρόγραμμά τη στη σωστή υλοποίηση τη οδηγία, αυξάνοντα και οργανώνοντα του ε, τακτικούς ελέγχους με την σύσταση εθνικών ομάδων εμπειρογνωμόνων. Ως προς την πρόληψη θα πρέπει να καλλιεργηθεί η νοοτροπία της πρόληψης της περιβαλλοντικής ζημιάς με μια εκστρατεία ενημέρωσης και τη δυνατότητα να προβλεφθούν ε, πρόστιμα οικονομικά ή άλλες μορφές, άλλες κυρώσεις για να ε, αναγκάζονται να λάβουν ευθύνη οι εταιρείε που είναι υπεύθυνε για περιπροδικές ζημιές. Μόνο έτσι μπορεί να εξασφαλιστεί η σωστή υλοποίηση τη οδηγία και η προστασία του περιβάλλοντο. Είμαι στη διάθεσή σα για παρατηρήσει, σχόλια και για να λάβω τι τροπολογίε σα τι ερχόμενε ημέρε. Ευχαριστούμε, κυρία Γκούτελαντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την εισηγητρία την κυρία Φεράρα για το σχέδιο έκθεσης είναι πολύ φιλόδοξο και ε, διεξοδικό. Έχοντας κατά νου ότι πέρασαν 13 χρόνια από την έγκριση του συστήματος για την παραγωγική ζημιά, ευτυχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύεται να θεωρήσει ως το δυνατόν συντομότερα. Γι' αυτό θα πρέπει να έχει ευρύ πεδίο η έκθεσή σας. Όπως σωστά είπε η κυρία Φεράρα στην έκθεσή της, είναι ιδιαίτερα προβληματική η υλοποίηση της ε, οδηγίας ELD για την παραγωγική ευθύνη από κάτω μέλος ή κάτω μέλος λόγω των διαφορετικών ε, τρόπων ερμηνείας και διαδικασίες για τα συγκεκριμένα όρια, ανώτατα όρια για να οριστεί η παραγωγική ζημιά. Είναι ένας από τους βασικούς φραγμούς για την ουσιαστική και πραγματική υλοποίηση της οδηγίας το πραγματικό ανώτατο όριο που μπορεί να καθορίσει την πραγματική ζημιά είναι πολύ ψηλό. Γι' αυτό θα προτείνω μια σχετική τροπολογία. Κατά τρίτο, είναι σημαντικό η έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να οριστεί η ζημιά και εις βάρος της ανθρώπινης υγείας και εις βάρος του περιβάλλοντος είναι καλό να συμπληρωθεί και το αναφέρω στην εισηγήτρια ότι χιλιάδες άνθρωποι χάνουν πρόημα τη ζωή τους λόγω της ατμοσφαιρικής ρήπανσης, κάτι που επίσης προκαλεί καρδιοαγγι... καρδιοαγγειακές παθήσεις. Όπως γνωρίζουμε, ε, με τα νέα επιστημονικά δεδομένα προκύπτει ότι η ατμοσφαιρική ρήπανση από βιομηχανικές δραστηριότητες και οι ευρωπαϊκοί κανόνες για τις εκπομπές των αυτοκινήτων ζημιώνουν την ε, κυριγία του κοινού, το περιβάλλον και δημιουργούν ε, ανισορροπίες σε επίπεδο βιολογικό και βιοεξελικτικό. Ξέρουμε υπό το φως σκανδάλων όπως το Dieselgate ότι πρέπει να αναλάβουμε δράση σχετικά. Ως και όδηση συγκήτρια για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες επί του θέματος ε, είμαι θερμά υπέρ μια έκκληση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, σκεφτεί την αναθεώρηση τη οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη πολύ σύντομα και να συμπεριλάβει και την περιβαλλοντική ζημιά που προκαλείται από ατμοσφαιρική ρήπανση, η οποία θα επιβαρύνει του αυτοκινητοπαραγωγού ε, με την σχετική προσαρμογή τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τι εκπομπέ των αυτοκινήτων. Μόνο εάν οι αυτοκινητοπαραγωγοί μπορούν να αναλάβουν ευθύνη για την ζημιά προκαλεί ατμοσφαιρική ρήπανση, τότε μόνο στο μέλλον η περιβαλλοντική ευθύνη και το σύστημα που καθορίζει θα μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να προλάβει την περιβαλλοντική ζημιά. Έτσι θα μπορούμε να υλοποιήσουμε σωστά την αρχή του «Οριπένων πληρώνει». Ευχαριστούμε. Δεν βλέπω άλλος κανείς να ζητά το λόγο. Η Επιτροπή. Από ό,τι φαίνεται όχι. Σε αυτή την περίπτωση, όντως η προθεσμία για την αποβολή των υπολογιών είναι 22 Ιουνίου, προφανώς 2017. Ωραία, θεωρούμε λοιπόν λήξαν το σημείο 8 και αν συγχωρείτε και συνεχίζουμε με το σημείο 8. Ανταλλαγή απόψεων για την αμοιβαία αναγνώριση της δέσμευσης και δίμευσης. Είμαι και σε αυτό το θέμα εισηγητής εγώ ίδιος. Να σας δώσω τις εξής πληροφορίες για το θέμα αυτό. Βάσει των προσφατότερων στοιχείων, οι παράτυπες αγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση φέρνουν 1% κέρδους, ε, από αναλογία ακριβώς το 1% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ για το 2010. Το να αποσπάσουμε τα κέρδη από τις εγκληματικές δραστηριότητες και να βεβαιωθούμε ότι το έγκλημα δεν φέρνει κέρδος είναι ο μόνος πραγματικά αποτελεσματικός μηχανισμός για να αντιμετωπίσουμε τις εγκληματικές ενέργειες. Η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που έχουν κερδιθεί με εγκληματικές δραστηριότητες στοχεύει να καταπολεμήσει και να αντιμετωπίσει το έγκλημα συμπεριλαμβανομένου του οργανωμένου, να αποζημιώσει τα θύματα και να προβλέψει πρόσθετους πόρους για να επενδυθούν ε, στις ε, διοκτικές δραστηριότητες ή άλλες πρωτοβουλίες για την πρόληψη του εγκλήματος. Ωστόσο, και παρόλο που υπάρχουσες στατιστικές είναι περιορισμένου χαρακτήρα, ο όγκος ε, ποσών που αυτή τη στιγμή ανακτώνται από τα κέρδη των εμπορικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια πολύ μικρή αναλογία. 98,9% του υπολογιζόμενου κέρδους από εγκληματικέ ε, δραστηριότητες δεν δημεύονται και παραμένουν στη διάθεση των εγκληματιών. Ένα εύρυθμο αρχείο για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων είναι προϋπόθεση για να δημεύονται τα εγκληματικά περιουσιακά στοιχεία, τα ε, περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με εγκληματικές δραστηριότητες. Και αυτό βεβαίως έχει να κάνει με την αμοιβαία αναγνώριση για την ε, δέσμευση και την δίμευση. Μετά την θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, η δίμευση έχει γίνει στρατηγική προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ένα ε, εργαλείο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος Η οδηγία 2014-42 προβλέπει κοινού ελέγχου κανόνε για την δέσμευση και δίμευση των ε, μέσων και ε, των ε, κερδών που προέρχονται από τι εγκληματικέ δραστηριότητε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν εγκρίθηκε η Οδηγία 2014-42, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε κοινή τους δήλωση κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξαναλέω, κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την αμοιβαία αναγνώριση της δέσμευσης και δίμευσης, καθώς και για τις ε, αποφάσεις σχετικώς, με την πρώτη δυνατή ευκαιρία, θεωρώντας την ανάγκη να υλοποιηθεί ένα σφαιρικό σύστημα για τη δέσμευση και την δίμευση των κερδών και των μέσων των εγκληματιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να προχωρήσει τωρινή πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μια απόκριση στις ε, εντοπισμένες ελλείψεις των υπαρχόντων εργαλείων για την αμοιβαία αναγνώριση και τις εκκλήσεις των συνομοθετών. Βασίζεται σε υπάρχουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αμοιβαία αναγνώριση της δέσμευσης και της δίμευσης και ε, ασχολείται με το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη έχουν αναπτύξει νέες μορφές δέσμευση και δίμευση των περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με το έγκλημα. Επίση, λαμβάνει υπόψη τι εξελίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο συμπεριλαμβανομένων των ελάχιστων προτύπων για την δέσμευση και την δίμευση, όπω προβλέπονται στην Οδηγία 2014 κάθετο 42. Ωστόσο, ενώ η οδηγία 2014-42 βελτιώνει τις εθνικές δυνατότητες να δεσμευτούν και να δημευθούν περιουσιακά στοιχεία, η τωρινή πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στόχο έχει να βελτιώσει την διασυνοριακή επιβολή των αποφάσεων για δέσμευση και δίμευση. Ως εκ τούτου, ο προτινόμενος κανονισμός έχει σκοπό να καλύψει όλες τις μορφές αμοιβαίας αναγνώρισης για όλες τις μορφές δίμευσης και δέσμευσης και των εντολών τους, των αποφάσεών τους, που εντάσσονται στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των εγκληματικών ε, ενεργειών. Μαζί με αυτές η ευρύτερη δίμευση ή δίμευση από τρίτο μέρος, η μη καταδίκη που βασίζεται σε ε, αποφάσεις δίμευσης. Ε, οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα προσεγγίσουμε την τωρινή πρόταση με συγκεκριμένε προτάσεις για να προσαρμοστούμε και να ευθυγραμμίσουμε την στάση μας σε αυτό το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτόν τον τομέα πολιτικής. Η κυρία Κάφμαν, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύντομα, Θεωρώ ότι πρόκειται πολύ σημαντικό θέμα και εσείς ο ίδιος ε, το αναφέρατε το νούμερο 110 δισεκατομμύρια τεράστιο ποσό ε, το οποίο τελικά μπορεί να χαθεί. Οπότε νομίζω πως ε, αξίζει να χαιρετήσουμε την προσπάθεια της Κομισιόν να απλοποιήσει εδώ το νομικό πλαίσιο. Θεωρώ ότι Παραδείγματο χάρη το να έχουμε τυποποιημένα έντυπα είναι πάρα πολύ σωστό. Αυτό το οποίο πρέπει να προσέξουμε είναι το θέμα του ποια άτομα αφορά. Πρέπει ακριβώς εδώ να προσέξουμε να μην υπάρχουν αδικαιολόγητες παρεμβάσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα και να έχουμε συντομότερες προθεσμίες οι οποίες όμως δεν θα είναι εις βάρος ε, της ε, εξέτασης ε, για το αν στα οικονομικά κάποια πράγματα. Τέλος, όσον αφορά τις οδηγίες ε, περί ανάκλησης θα πρέπει νομίζω να έχουν προβάδισμα ή απαιτήσει ε, των θυμάτων έναντι των υπολείπων. Αυτά ε, ως προς την πρόταση της Κομισιόν, την οποία σε γενικές γραμμές εμείς υποστηρίζουμε. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα, κυρία Κάφμαν, να σας ρωτήσω τι εννοούσατε ε, όταν είπατε για προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, μια πρόταση παραπάνω μπορείτε να μας πείτε. Ακούστε, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι πρέπει να προσέξουμε να μην υπάρξουν δικαιολόγητες επιθέσεις ε, σε βάρος προσώπων να μην υπάρξει αδικία. Αυτό είπα ότι πρέπει να προσέξουμε. Yes, of Thank you. Βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω να θέλει κάποιος να στο λόγο. Επομένως, μπορούμε να ολοκληρώσουμε το σημείο αυτό της μέσης διάταξης και να συνεχίσουμε με το σημείο 9 που είναι εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης για το σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και κατά τις οδηγίες 2058, κύριος Φως που είναι ο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως και με την ανταλλαγή απόψεων Εγώ ασχολούμαι με την πρόταση e-privacy της Κομισιόν και έχω να εκφράσω τη δυσαρέσκειά μου με αυτή την πρόταση σε ό,τι αφορά τους στόχους δηλαδή που θέλουμε να εφαρμόσουμε για την ψηφιακή αγορά και τα λοιπά, αυτούς δεν μπορούμε να τους πετύχουμε. Ίσα ίσα πηγαίνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση πολλές από τις διατάξεις ε, της πρότασης της Κομισιόν και επίσης υπάρχουν πολλά επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία μπορούμε πλέον να εφαρμόσουμε κατά την άποψή μου. Επίσης όλα αυτά οδηγούν σε μία συνέπεια με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και σε αντιφάσεις και άρα δημιουργείται μεγάλη ανασφάλεια δικαίου ό,τι αφορά την ε, διαχείριση δεδομένων. Και παράλογες ε, τελικά είναι οι επιπτώσεις όταν αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό που θα προτιμούσα εγώ θα ήταν η όλη πρόταση να διαγραφεί και να βάλουμε μόνο μια πρόταση που να γίνεται λόγος για το απόρριτο της, της επικοινωνίας. Αυτό νομίζω ότι θα αρκούσε. Αυτό που προσπαθούμε τώρα να κάνουμε, κατά την άποψή μου τουλάχιστον, ε, μπορούμε να προσπαθήσουμε να, το, να πάμε αυτή την πρόταση με διάφορες διορθώσεις και τροπολογίες προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν νομίζω ότι αλλάζει και τίποτα ουσιαστικά. Σίγουρα αυτό που θα χρειαζόταν θα ήταν περισσότερο θάρρος και δημιουργικότητα και όχι να παραμένουμε ε, κολλημένοι σε παλές δομές, ε, γιατί θέλουμε να πετύχουμε αυτή την ψηφιακή επανάσταση και δεν το πετυχαίνουμε αυτόν τον τρόπο. Αν δει κανεί ε, ε, τον ειδικό αυτό που θέλει για το e-privacy να είναι αυτό ο κανονισμό της Κομισιόν, αυτό το λέξη specialis, εγώ διερωτώ. Γιατί έχει κάτι κακό ο γενικό κανονισμό προστασία Δεδομένων, δεν θα μπορούσε δηλαδή να ενταχθεί αυτό το στοιχείο στον κανονισμό, να πούμε δηλαδή τι ε, χρειάζεται να προσθεθεί, δηλαδή το απόρριτο ε, της επικοινωνίας. Κατά την άποψή μου αυτό θα ήταν αρκετό, πολλοί λένε βέβαια. Αυτό δεν χρειάζεται καν να γίνει γιατί έχουμε τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων που είναι αρκετή ε, νομική βάση αυτά, αλλά τέλο πάντων. Αν έχουμε την επεξεργασία δεδομένων χωριστά από την επικοινωνία, θα χρειαζόταν να αναφέρουμε εδώ σε ό,τι αφορά το απόρριτο μόνο την επικοινωνία. Επίση υπάρχουν ε, παράλληλε δομές με τον κανονισμό. Με τη δική μου έκθεση εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω είναι να οδηγήσω τις διατάξεις προς μια πιο σωστή κατεύθυνση. Δεν ξέρω αν έχω καλύψει όλα τα όσα έχω θεωρήσει σημεία που χρήζουν κριτικής. Αυτό που λείπει Να δούμε και τα γενικά και τα ειδικά, ε, θα σας δώσω κάποια παραδείγματα. Στο άρθρο 4, για παράδειγμα, έχουμε τον κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Δεν ε, τηρείται ο κώδικας ε, με αυτό το άρθρο. Τον παραβιάζει. Πριν την συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κώδικα θα έπρεπε να εφαρμοζόταν ε, αυτός ο κανονισμός. Αυτό είναι συστημικό λάθος και πρέπει να το διορθώσουμε. Είπα για τον κανονισμό, τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, ποια είναι τα όρια, δεν είναι σαφή και θα έπρεπε να το ξεκαθαρίσουμε καλύτερα. Να δούμε δηλαδή τι είναι λογική συνέπεια και να ε, καταργήσουμε, να απαλείψουμε τις ασυνέπειες. σε ό,τι αυτά τα μεταδεδομένα, για παράδειγμα, και την προστασία των δεδομένων, να γίνονται ε, κάποιες, μάλλον προκύπτουν κάποιες παράλογες επιπτώσεις και συνέπειες. Αυτά τα όρια, όπως είπα, μεταξύ απόρριτου της επικοινωνίας και επεξεργασίας δεδομένων. με συμμετοχή των συνδεδεμένων συσκευών και μηχανών. Και εδώ πάλι μπορεί να προκύψουν κάποιες παράλογες ε, και μη δυνατόν να προβλεφθούν εκ των προτέρων ε, συνέπειες όταν έχουμε αυτές, αυτή την επικοινωνία μηχανής, μηχανής θα μπορούσε ε, να λειτουργήσει πολύ καλά και να συνδεθεί, μάλλον να περιληφθεί η επικοινωνία μηχανής μηχανής, αλλά τι θα γίνει η συγκατάθεση με τη συγκατάθεση στην επικοινωνία μηχανής μηχανής. Γιατί μέχρι στιγμής προβλέπεται μόνο η συγκατάθεση ανθρώπων, όχι μηχανών. Άρα θα προκύψουν διαφορές στο σύστημα. Επίσης, τι γίνεται με την επεξεργασία ανωνύμων δεδομένων και τι θα γίνει με τη συγκατάθεση. Και αυτό δεν είναι λογικό, όπως προβλέπετε. Πώς μπορώ να επεξεργαστώ ανώνυμα δεδομένα. Υπάρχει επίσης μια πρόταση για τα, για τα cookies. Κατ' εμέ αυτή η ρύθμιση ε, κάνει αυτό που δεν θέλουμε, δηλαδή από τις μεγάλες επιχειρήσεις, εμείς θέλουμε περισσότερο ανταγωνισμό, αλλά το αντίθετο ε, δημιουργείται εδώ. Επίσης, ό,τι αφορά το άρθρο 5, το ε, email τίθεται σε κίνδυνο με, τη διαδικασία, με την διατύπωση. Η ίδια η υπόσταση του οικονομικού ταχυδρομικού υποαφισβήτηση με αυτή τη διατύπωση. Προβλήματα λοιπόν υπάρχουν με την εφαρμογή. Η ερώτηση είναι κατά πόσον δηλαδή χρειάζεται αυτή η πρόταση, αν είναι κάτι θετικό που θα μας πάει μπροστά για να πετύχουμε την ψηφιακή αγορά. Δυστυχώς λείπουν πάρα πολλά και εγώ είμαι άκρο δυσαρεστημένος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία εκπροσωπείται σήμερα εδώ και ίσως θα μπορούσε να τοποθετηθεί για μια ακόμη φορά πάνω σε αυτά. Πραγματικά μου είναι πολύ δύσκολο να βρω κάτι θετικό ε, σε αυτή τη λογική μιας νομοθετικής πρότασης. Φυσικά και θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, αξιοπιστία Θέλουμε να έχουμε τη νομική βάση για την προστασία των δεδομένων. Αλλά έτσι όπως έχει διατυπωθεί αυτή η πρόταση, περιλαμβάνει πιο πολλά μειονεκτήματα από ό,τι πλεονεκτήματα. Και κατά την άποψή μου πρέπει αυτό να αλλάξει. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Ντελβό. Sorry, Mr. Lode. Ε, κύριε Σοντέ. Ναι, ναι. Εγώ προσωπώ την Άλντε Πρώτα απ' όλα λοιπόν να ευχαριστήσω τον κύριο Φως για τη δουλειά που έχει κάνει και ειδικά για τα λόγια που είπε. Επί της αρχής συμφωνώ πλήρως. Δεν θα ήθελα επίσης ε, να αμφισβητήσω και εγώ τη Γενική Οδηγία Προστασίας ε, Προσωπικών Δομένων ή να δημιουργηθούν εδώ πέρα διπλές ε, δομές. Και πρέπει να προσέξουμε να μην υπάρχει κάποια αντίφαση εδώ σε σχέση με το e-privacy. Αλλά έχουμε δυστυχώς ε, πολύ λίγο χρόνο γιατί η μετάφραση ήρθε σήμερα το μεσημέρι μόνο. Εντάξει, εγώ δεν είχα πρόβλημα, αλλά Πρέπει όλοι οι βουλευτές ε, να έχουν ε, τις ίδιες ε, δυνατότητες. Πρέπει λοιπόν την Πέμπτη εδώ να προσέξουμε να, ότι έχουν όλοι τη δυνατότητα και να πω ότι χρειάζεται λίγος χρόνος για να δούμε και τις τροπολογίες Κατά τα λοιπά, συμφωνώ απολύτως με την προσέγγιση του κυρίου Φως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Ντελβό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ως προς το ότι είναι άκρος πολύπλοκη αυτή η πρόταση. Και εγώ προσπαθώ να καταλάβω ε, και να βρω μια άκρη με τους διάφορους κανονισμούς και οδείς και δεν είναι προφανές. Λοιπόν, άρα, χρειάζεται ένας κανονισμός για το απόρριτο. Του περιεχομένου το απόρριτο. Και νομίζω από αυτό συμφωνούμε όλοι. Αλλά από εκεί και πέρα. Δυσκολεύομαι τα μάλλα με τους ορισμούς. Μιλάμε για δεδομένα. Και μετά για με, μεταδεδομένα. Εγώ εντάξει, μπορώ να καταλάβω ποια είναι η διαφορά γιατί τα δεδομένα τη χάνουν προστασία στο πλαίσιο του Γενικού Ενωσμού και τα μεταδεδομένα δεν ρυθμίζονται. Τα δεδομένα, αυτά το τα μεταδεδομένα δηλαδή, είναι εμπιστευτικά, είναι απόρριτα. Αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ προσωπικά. Θα ήθελα λοιπόν να το συζητήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος. Ε, Συμφωνώ με την ανησυχία του εισηγητή για τους ορισμούς, γιατί υπάρχουν παραπομπές στο Γενικό Κανονισμό προς Δεδομένων, αλλά και στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ελεκτρονικών Επικοινωνών, που εξ όσων γνωρίζω θα αλλάξει σύντομα. Άρα, ποιον ορισμό θα επιλέξουμε και τι συμβατότητα και συνέπεια θα υπάρχει μεταξύ τους ορισμούς και τα διαφορετικά κείμενα. Τώρα, επί της αρχής, πρώτο μας μέλημα είναι η μεγαλύτερη δυνατή προστασία του περιεχομένου και εδώ στρέφουμε στους πραγματικούς ειδικούς στο γενικό κανονισμό υπάρχει έννοια του θεμητού συμφέροντος. όχι για παραβιωστό του απορρίτου, αλλά το αν υπάρχει νόμιμο συμφέρον μπορούν να το παραβιάσουν το απόρριτο αν θέλετε. Άλλο τα δεδομένα όμως και άλλο το περιεχόμενο. Πού υπάρχει νόμιμο συμφέρον για το περιεχόμενο. Δεν το βλέπω μόνο αν το ζητήσει ο χρήστη. Αν θέλει δηλαδή να έχει μια μετάφραση. Τηλεφωνικά. Από εντάξει, αυτό σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να ακούσει το περιεχόμενο γιατί αλλιώς δεν μπορεί να γίνει η μετάφραση. Επίσης θα ήθελα να υπάρχει πρόταση και έλεγχος για τους ανηλίκους, για τα παιδιά. Ίσως χρειάζεται να ελέγχονται οι συνομιλίες τους. Αυτό κατ' δεν, ε, από ό,τι ξέρω δηλαδή, δεν υπάρχει στο γενικό κανονισμό, άρα και αυτό το θέμα νομίζω ότι πρέπει να ε, το δούμε σε βάθος. Δεύτερη ε, ανησυχία μου, που το είπε και ο κύριος Φως, αλλά δεν ξέρω πώς μπορούμε να το λύσουμε το πρόβλημα, είναι να μην ευνοούμε μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις, τα cookies, σε αυτή την επιλογή. Επίσης, νομίζω ότι η συγκατάθεση πρέπει να αφαιθεί για τον πελάτη. Ξέρω ότι είναι πολύ κουραστικό να πατά συνέχεια ένα κουμπί και κάποιες φορές ή τις περισσότερες δεν διαβάζουμε καν που δίνουν τη συγκατάθεση. Θα έλεγα λοιπόν να δίνετε μια εύληπτη εξήγηση στο χρήστη αλλά παρόλα αυτό ο Χρήστος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να πει όχι. Ναι ή όχι τέλο πάντων να πει. Μπορεί να μην τα διαβάζουν πολύ, αλλά για κάποιους είναι πάρα πολύ σημαντικό και γιατί να το καταργήσουμε, δεν βλέπω το λόγο. Αυτές είναι οι πρώτες μου σκέψεις. Έχουμε δρόμο μπροστά μας ακόμα. Για να καταλήξουμε σε μία γνωμοδότηση. Επίσης, το λέω από τώρα, δυστυχώς δεν θα είμαι διαθέσιμη για μια συνεδρία σε σκιωδών εισηγητών. Λυπάμαι πολύ. Άρα θα ήθελα να δω κάτι δίαν, ε, να κλείσω ένα ραντεβού ιδιωτικό με τον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριο Άντερσον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για την έκθεσή του. Επιτέλους μπορώ να διαβάσω σε μια γλώσσα που καταλαβαίνω. Και έχω αρχίσει σιγά έτσι να ασχολούμαι με το θέμα. Πρώτα, παρατηρώ ότι ο εισηγητής ε, είναι πολύ επικριτικός για το άρθρο 4 το άρθρο 4 όμως είναι ένα από τα λίγα άρθρα που δεν προτείνει να αλλάξουν. Νομίζω λοιπόν πως θα μπορούσε να ξεκαθαρίσει τις ε, απόψεις του αυτές ε, και θα του ήμουν ευγνώμων. Σε σχέση με τα όσα υπόθηκαν για το άρθρο 5 που λέει ότι απειλεί την ε, ύπαρξη του email. κατάλαβα πώς ε, γίνεται αυτό. Οπότε θα ήθελα μια εξήγηση. Τώρα, σε κάπως πιο γενικά ζητήματα, δεν κατάλαβα καλά την βασική κατεύθυνση Μάλλον δεν του αρέσει αυτή η πρόταση και προσπαθεί να διαγράψει πολλά πράγματα. Φαίνεται ότι θέλει να ευνοήσει τα συμφέροντα των επιχειρήσεων στο μέτρο του δυνατού και να διευκολύνει τις εταιρείε να συλλέξουν πληροφορίες για τους πελάτες τους. Οι πράσινοι από την άλλη θα θέλαμε να ενισχύσουμε την ιδιωτικότητα και την ακαιρεότητα των πολιτών και θα πάμε κυρίως προς την άλλη κατεύθυνση. Προτιμούμε την πρόταση της Κομισιόν προβλέπω ότι θα έχουμε κάποιες συζητήσεις και αναρωτιέμαι εάν θα έχει αρκετό χρόνο η Επιτροπή να ψηφίσει πριν την Λίμπη γιατί θα έχουμε μία μέρα μόνο πριν ψηφίσει η Λίμπη είναι πρόβλημα αυτό Και τώρα παίρναμε σε κάποια άλλα ζητήματα. Εγώ προτιμώ την διατύπωση της Κομισιόν για το άρθρο 1 και βασικά προτιμούμε την προσέγγιση την συνενετική. Δηλαδή η επεξεργασία των μεταδεδομένων θα πρέπει να βασίζεται στην συνένεση. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε κατεύθυνση, να φύγουν οι αναφορές για την παρακολούθηση cookies κτλ. Και γενικά είμαστε υπέρ της ε, στεναρούς, ε, της στεναρής ε, προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Επίσης, θέλαμε να υπάρξει απαγόρευση της παρακολούθησης ε, στο διαδίκτυο μέσω Bluetooth ή Wi-Fi και θεωρούμε ότι θα πρέπει η ιδιωτικότητα από τη φάση του σχεδιασμού να περιληφθεί ως σημαντική αρχή σε αυτόν τον κανονισμό. Επίσης, η απευθείας διαφήμιση θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο εάν το έχει επιτρέψει ο τελικός χρήστης. Ελπίζω λοιπόν να συμφωνήσει με όλα αυτά ο εισηγητής. Σας ευχαριστώ. Η Κομισιόν θέλει τον λόγο. Έχουμε την κυρία Σπανού από την Γενική Διεύθυνση Connect. Ναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ακριβώ να έτσι λέγομαι. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Φω, όλο ιδιαίτερο για την ομοδότηση. Εδώ είμαστε να προσπαθήσουμε να διαλευκάνουμε κάποια ζητήματα. Ακούσαμε ότι και συμφώνησατε όλοι ότι είναι πολύπλοκη η πρόταση και νομίζω ότι αυτή είναι η γενική προσέγγιση. Δεν είναι και τόσο ε, μεγάλη υποστήριξη της Επιτροπής σας από τη Θέλω να συνεργαστούμε όσο μπορούμε. Θα έρθουμε και στη συνεδρίαση των σκιωδών, μας ε, προσκαλέσατε και θα τα δούμε από κοντά. Ο ε, όλος στόχος είναι μεγαλύτερη προστασία Ε, σε σχέση και με τους, ε, τις διατάξεις που πρέπει ο γενικός κανονισμός ε, και διευρύνουμε έτσι το πεδίο εφαρμογή των κανόνων που ισχύουν για τις παραδοσιακές τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις τα λεγόμενα over the top καλύπτονται δηλαδή επιφύης επιχειρήσεις και πρέπει να σας πω ότι έχουμε μια οδηγία για την ηλεκτρονική προστασία τη ιδιωτικότητα. Δεν ξεκινάμε από το μηδενό. Προσθέτουμε αυτό το κομμάτι στο πεδίο γιατί γνωρίζουμε ότι οι καταναλωτέ όλο και περισσότερο χρησιμοποιούν αυτέ τι νέε υπηρεσίε και ανησυχούν ιδιαίτερα για τη χρήση των δεδομένων του. Ε, και ε, έχουμε προτείνει κανονισμό αντί οδηγία ακριβώς γιατί πιστεύουμε ότι έτσι θα υπάρχει νομική ασφάλεια για χρήστε και επιχειρήσει. Η ιδιαιτερότητα και έρχομαι ε, στο privacy ε, και για τα δεδομένα και για τα μεταδεδομένα. Τι εννοώ με τα δεδομένα, το χρόνο μιας κλήσης, ε, το τόπο, επειδή είναι ευαίσθητα αυτά τα δεδομένα. Αν ο χρήστη δεν δώσει τη συγκαταθεσή του, τότε τα δεδομένα είτε θα πρέπει να νομιμοποιηθούν, να διαγραφούν, εκτό αν είναι απαραίτητα για την τιμολόγηση. Για παράδειγμα, όταν δοθεί συγκατάθεση για, τη, για τα δεδομένα επικοινωνιακά, είτε είναι με τα δεδομένα, είτε είναι περιεχόμενο για την επεξεργασία του, οι παραδοσιακέ επιχειρήσει θα μπορούν να παράσχουν παραδοσιακέ πληροφο... υπηρεσίε. Θέλουμε δηλαδή μια αγορά που όλοι να δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να να υπάρχουν ε, κάποιοι χάρτες, heat maps, θα μπορούν να βοηθήσουν. Allowing people Σε ό,τι αφορά τους κανόνες για τα cookies, θέλουμε να έχουμε κάτι που να μπορεί να είναι πιο φιλικό για το χρήστη. Αυτό που χρειάζεται να διευκρινιστεί ίσως είναι. Σε ποιον εφαρμόζονται οι κανόνες. Σε όλους όχι στους μεγάλες επιχειρήσεις και στις μικρές επιχειρήσεις στην αγορά. Δεν υπάρχει διάκριση. Αυτό που θέλαμε ήταν να έχουμε απλά ρυθμίσεις ε, στο browser. Πάλι να υπάρχει έλεγχος από το χρήστη. Που μπορεί να αρνηθεί τα cookies και άλλα αναγνωριστικά. Αν όμως βελτιώνουν κάποια cookies στην εμπειρία της ε, περί διάβασης του διαδικτύου δεν χρειάζεται να υπάρξει συγκατάθεση αυτά τα συγκεκριμένα κούκς αφόσον δεν ε, παρεμβαίνουν ε, στα προγράμματα. Άρα διευκρινίζουμε ότι μπορεί να υπάρχουν επιπτώσεις που δεν χρειάζεται και να δοθεί συγκατάθεση. Γιατί δεν έχει να κάνει με την προστασία της επικοινωνίας, ε, του απορρίτου, της επικοινωνίας κτλ. Ένα άλλο θέμα που είδαμε ότι υπάρχει μια πρόταση διαγραφής είναι η Direct Marketing Communications, άμεσες, ε, άμεση επικοινωνία για στόχους marketing. Ακούστε, η πρόταση για email, SMS μιλάμε τώρα, ή αυτοματές συσκευές. Αν δεν δοθεί συγκατάθεση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. είτε προστατεύονται εξ ορισμού, αλλά ανάλογα με την νομοθεσία της κάθε χώρας. Είτε δεν δέχονται κλήσεις ε, marketing, σκοπούς marketing. Έτσι εξελίσσονται οι κανόνες. Και δεν ξέρω γιατί προτείνεται να διαγραφούν. Σε ό,τι αφορά τους ορισμούς. Όταν κάναμε την πρόταση, θέλαμε να ευθυγραμμιστεί με δύο μέσα. Το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων που έχει εγκριθεί και δεύτερον, πράγματι τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ελεκτρονικών Επικοινωνίων. Για να έχουμε αυτή την ασφάλεια δικαίου. Η πρόταση σε αυτόν τον κώδικα, τον Ευρωπαϊκό, συζητείται και επειδή είναι παράλληλοι, νομίζω θα εγκριθούν περίπου ταυτόχρονα για να δημιουργηθεί ασφάλεια δικαίου. Δεν το έχουμε παραβλέψει αυτό το στοιχείο, το αντίθετο. Προσπαθούμε να υπάρξει αυθυγράμμιση και με το Γενικό Κανονισμό αλλά και με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα. Ελπίζω αυτοί οι μικρές διευκρινήσεις να σας βοήθησαν. Φυσικά μόλις διαβάσαμε την έκθεση, αλλά είμαστε στη διάθεσή σας να συνεργαστούμε και περαιτέρω και να σας δώσουμε όποια διευκρίνηση χρειάζεται. Πρόεδρος, δεν ξέρω αν θέλει να απαντήσει ο κύριος Φως πριν δώσω τον λόγο μου στον κύριο Φώσα. Θα σας διακόψω όταν ήρθε ο κύριος Άνση, αν δεν το ολοκληρώσει κύριε Φως. Κύριο Φω, ναι, σε αυτά τα δεδομένα. Κατά την άποψή μου τα δεδομένα είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατ' εμέ. Με ποιον μιλάμε, πόση ώρα μιλάμε, από πού καλούμε, προ τα πού κτλ. Άρα για μένα είναι καθαρά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Σε ό,τι αφορά την σχέση με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα και το αν υπάρχει συμβατότητα και συνέπεια. Πράγματι, εγώ θεωρώ ότι αυτό πρέπει να συμβεί. Στο 4, για το άρθρο 4, Σε ό,τι αφορά τον Ευρωπαϊκό, Ευρωπαϊκό, Κώδικα, σε ό,τι αφορά την προθεσμία ε, εφαρμογής, το αναφέρω ότι πρέπει να γίνει παράλληλα η έγκριση ή τέλο πάντων η χρήση του κανονισμού αυτού, του κώδικα αυτού μαζί με το γενικό κανονισμό. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στο άρθρο 4. Η αλλαγή πηγαίνει, αφορά την προθεσμία, τον χρόνο έναξης ισχύω εφαρμογής. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 5, και αυτό είναι ενδιαφέρον, για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, για το email. Βέβαια είναι και θέμα ερμηνεία. Πώς ερμηνεύουμε αυτά τα μεμονωμένα ζητήματα. Σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρονικά δεδομένα, υποκλοπή, ε, αποθηκεύση παρακολούθηση κτλ. για να μην υπάρξει επίθεση, θα πρέπει να πάψει αυτή η επικοινότητα στο μότερο δυνατό. Τι γίνεται, δηλαδή το email πηγαίνει από τον Α στον Β και μετά σβήνεται, διαγράφεται για να μην μπορέσει να έχει πρόσβαση κάποιο τρίτο. Θα πρέπει να δούμε αυτό τι επιπτώσει μπορεί να έχει όμω. Ε, αν η διατύπωση είναι σαφή τελικά και νόμιμη, νομικά σωστή. Επίσης, ένα συνεπές δίκαιο. Για τον νόμο συμφέρον που, που είπατε, ναι. Το θέμα είναι η ασφάλεια δικαίου και η σαφήνεια. Θα πρέπει να είναι σαφές και για τους χρήστες αλλά δυστυχώς δεν είναι καθόλου ξεκάθαρες οι διατάξει σχέση και με το Γενικό Κανονισμό Προστασία Δεδομένων. Θα πρέπει να το προσέξουμε λοιπόν για τις μικρές μεγάλες επιχειρήσεις. Ακούσαμε τι είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, φυσικά αυτό ο κανονισμό ισχύει και για τι μικρέ και για τι μεγάλε επιχειρήσει. Εγώ μιλάω για τι επιπτώσει. Ότι οι μεγάλε επιχειρήσει ε, δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα και μπορούν να φέρουν σε πέρα όλα όσα ζητούνται εδώ. Όχι όμω οι μικρέ επιχειρήσει. Γι' αυτό λέω ότι σε ό,τι αφορά τα cookies, ε, ουσιαστικά ε, ευνοούνται οι μεγάλες επιχείρησεις, κάτι το οποίο δεν θα θέλαμε. Και σε ό,τι αφορά τη συγκατάθεση, αυτή η εστίαση στην ε, συγκατάθεση νομίζω ότι αδικά θα καταργήσει την προστασία της ιδιωτικότητας, ε, διότι όλοι μπορεί να ε, εγκρίνουμε και να συγκατατιθέμεθα σε οτιδήποτε αδιακρίτως. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει κάποια άλλη δυνατότητα σε ό,τι αφορά τη συγκατάθεση. γιατί πολλές φορές τη δίνουμε έτσι τη συγκατάθεση. Το θέμα είναι να έχουμε διαφάνεια, κυριαρχία δεδομένων, ε, τις εξαιρέσεις, τις ε, αντιτάξεις, αυτοεξαίρεση, αντίταξη, όλα αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα δούμε. Όλα αυτά όμως είναι πιο ε, σίγουρα από το να δίνουμε, να πατάμε το κουμπί ναι, ναι, ναι στη συγκατάθεση χωρίς να διαβάζουμε καθόλου τι λέει το κείμενο πριν το πατήσουμε αυτό το κουμπί. Ευχαριστώ. 29 Ιουνίου είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες. Είναι έτσι. Έτσι φαίνεται. Ευχαριστώ. Θα ζητήσω από τον κύριο Τζαμπάσκι και την κυρία Ντελβό αν μπορούμε να αναβάλουμε τα σημεία τους για αύριο μετά τις ψηφοφορίες. Αύριο μετά τις ψηφοφορίες, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Καλωσορίζω τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Άνσιπ, στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, ξανά, στα πλαίσια του διορθωμένου διαλόγου μεταξύ των θεσμικών οργάνων και χωρίς ε, καθυστερήσεις να δώσω τον ε, λόγο στον Επίτροπο. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Πριν δύο χρόνια ξεκινήσει η στρατηγική της ψηφιακής αγοράς και στα πλαίσια αυτής έχουμε ετοιμάσει 35 προτάσεις, εκ των οποίων 21 νομοθετικές. Είναι μεγάλη μου ικανοποίηση να μπορώ να πω ότι χάρη και στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων πετύχαμε να τις φέρουμε σε αίσιο πέρας με συνένεση. Μιλάω για την κατάργηση των τελών roaming, της περιαγωγής, θέμα που συζητήθηκε τελευταία φορά την περασμένη εβδομάδα, ένα τεράστιο επίτευγμα για όλους τους πολίτες μας. Επίσης τα 700 MHz και το σχετικό φάσμα που επέτρεψε το 5G να γίνει μια άμεση πραγματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζουμε να πετύχουμε και εδώ συμφωνία. Επίσης το Wi-Fi for you, θέματα και φάκελοι που έχει εξετάσει και η Επιτροπή Γιούρι. Επίσης και σε άλλα αποτελέσματα είχατε μεγάλη επίδραση όπως την ε, φορητότητα και εκεί πετύχαμε συμφωνία και του χρόνου ο κόσμος δεν θα, πρέπει, δεν θα πια να πληρώνει αυτές τις υψηλές τιμές περιαγωγής και θα χρησιμοποιεί πολύ περισσότερο τις δυνατότητες ε, του διαδικτύου όταν θα ταξιδεύει ε, και θα θέλει τον ε, ψηφιακό του περιεχόμενο και σε μια άλλη χώρα. Συνδίκη του Μαρακές. Χάρη στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, οι τυφλοί θα έχουν πολύ περισσότερη πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο. Πολύ σημαντικό για όλους τους τυφλούς πραγματικές επιτυχίες και τώρα έχουμε φτάσει σε μια φάση όπου πολλές από τις προτάσεις αυτές είναι έτοιμες για την τελική φάση λήψης απόφασης. Αναμένω λοιπόν την επικοδηματική μας συνεργασία με την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων για όλα αυτά τα θέματα. Τον Μάιο ξεκινήσαμε τη στρατηγική για την ενιαία ψηφιακή αγορά για να εντοπίσουμε νέους τομείς όπου έπρεπε να δώσουμε πολύ περισσότερη προσοχή στο τι συμβαίνει. Και όπως ξέρετε μιλάω για τις επιγραμμικές πλατφόρμες που είναι ένα θέμα που συχνά ανακύπτει. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ε, μη ικανοποιημένες, ανικανοποίητες. Προσπαθούμε να ε, προσαφηνίσουμε λοιπόν ε, την διασύνδεση του θέματος αυτού με τις επιχειρηματικές πρακτικές και να δούμε και τι θα επιφέρει στην πραγματικότητα το Brexit, διότι πολλές χώρες ε, περνάνε τους δικούς τους νόμους, ε, έχουν δικούς τους νόμους αντιμετώπισης των εκφράσεων μίσους, ε, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και άλλα κράτη-μέλη τα σκέφτονται αυτά και τους απασχολούν. Στόχος μας λοιπόν είναι να έχουμε μεγαλύτερη σαφήνεια. Ταυτόχρονα όμως θέλουμε να προστατεύσουμε και τις αρχές του ηλεκτρονικού εμπορίου όπως καταγράφονται στην οδηγία αυτή για την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία λόγου. Δεν θέλουμε να αγγιχθεί η αρχή του ασφαλούς λιμένα, όπως προβλέπεται από την οδηγία. Κατά δεύτερον, χρειάστηκε να ασχοληθούμε με το θέμα της ψηφιακής οικονομίας καθώς 21 ε, κράτη-μέλη είχαν ε, σχετική νομοθεσία για τον ε, γεωγραφικό εντοπισμό των δεδομένων. Είναι κάτι ιδιαίτερα δαπανηρό και εμποδίζει τη δημιουργία νέα αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτο κλάδο όπου δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή ήταν η κυβερνοασφάλεια. Ξεκινήσαμε τη στρατηγική κυβερνοασφάλεια το έτος 2013 και μπορούμε να πούμε ότι δεν πέρασαν και πολλά χρόνια από τότε που ε, λειτουργεί αυτή η στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κυβερνοασφάλεια, αλλά μπορούμε ήδη να πούμε ότι οι κυβερνοαγκληματίες ε, έχουν κάπως συμμαζευτεί. Καθώς ε, με το διαδίκτυο των πραγμάτων, το Internet of Things, είχαμε άλλα δεδομένα τότε που εγκρίθηκε η στρατηγική, όμως με τι διασυνδεδεμένε διασυνδεδεμένες μάλλον και τα ενδεχόμενα μαζικών επιθέσεων, δίντος, πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη μας διαφορετικά την κυκλοφορία των δεδομένων και να πάρουμε πολύ πιο σοβαρά υπόψη την κυβερνοασφάλεια, ιδίως όταν χρειάστηκε να συμφωνήσουμε διεθνώς κοινά ε, πρότυπα κυβερνοασφάλειας για το διαδίκτυο των πραγμάτων. Υπάρχει και ηλεκτρονική υγιεινή. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι πριν φάμε πρέπει να πλύνουμε τα χέρια μας, αλλά όταν μιλάμε για την κυβερνοασφάλεια κάποιος άλλος πρέπει να τα πλύνει. Ε, είναι γνωστό αυτό το επεισόδιο με τον Υπουργό Εξωτερικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά εάν δούμε τα δεδομένα, μπορούμε να περιορίσουμε κατά το 80% της επιθέσεις DDoS, αρκεί ο κόσμος να λάβει υπόψη του σοβαρά τα δεδομένα της ασφάλειας και να αλλάξει κάποιες φορές τα default, τις default ρυθμίσεις της ασφάλειας που πρέπει κανείς να της προσωποποίηση. Όταν αγοράζει κανείς μια ηλεκτρική σκούπα, ας πούμε, ή ένα ρομπότ που κουρεύει το γρασίδι, δεν φοβάται κανείς. Όμως, όταν φοβάται με του το κλέψουνε το ρομπότ που έχει έξω στον κήπο γιατί με αυτό κουρεύει το γρασίδι, εκεί μπορεί και να αλλάξει τα δεδομένα ασφάλειας. Έτσι πρέπει να σκεφτεί ο κόσμος. Επίσης πρέπει να δούμε τις, ε, τα σημεία συμφόρησης ε, χάρη στη, που οφείλονται στις διασυνδεδεμένες συσκευές. Πρέπει να δούμε τις επιχειρησιακές λειτουργίες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης 21-24-7 και να δούμε πόσο τα κράτη-μέλη μπορούν να συνεργαστούν με τις Βρυξέλλες, την Europol επίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε 30 ανθρώπους να εργάζονται για τα θέματα αυτά, αλλά 30 άτομα δεν είναι καν αρκετά. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε καν ήδη τις 27 τις 7-24 ε, ε, υπηρεσίες. Ξέρουμε λοιπόν ότι η ελευθερία είναι αναγκαία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ξέρουμε επίσης ότι μόνο σε 5 τρίτα των κρατών μελών υπάρχουν επιχειρησιακές δυνατότητες. Πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί για την κυβερνοασφάλεια και τα σχετικά στοιχεία. Τώρα να αναφέρω μερικά θέματα ιδιαίτερο ενδιαφέροντος. Η προτινόμενη οδηγία για τα δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία και την ενιαία ψηφιακή αγορά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα φιλόδοξο βήμα για να προάγουμε την πολιτιστική πολυφωνία, την πρόσβαση προς και την προστασία του ψηφιακού περιβάλλοντος. Εδώ προβλέπονται επικαιροποιημένοι και σύγχρονοι κανόνες για όλους τους φορείς της αγοράς. Νομίζω ότι έχουμε πετύχει καλό σημείο ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων των χρηστών του διαδικτύου, των κατόχων των δικαιωματογνωτικής ιδιοκτησία και των παρόχων υπηρεσιών, ώστε να έχουμε λύσεις αγοραστραφής, οι οποίες να επιτρέψουν οι χρήστες να είναι εκ των προτέρων προστατευμένοι. Να καλέσω την Επιτροπή σας να διατηρήσει αυτό το καλό σημείο της Ευρωπίας. Επίσης, θεωρώ ότι πρέπει να επιστήσω την προσοχή σας σε τουλάχιστον μερικά θέματα. Το πρώτο θέμα έχει να κάνει με τις εξαιρέσεις στα δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησίας, ιδιαιτέρως ε, τα κείμενα και την ε, άντληση κειμένων. Η κάτοχοι αυτής της εξαίρεσης θα πρέπει να είναι μόνο ερευνητικά ιδρύματα, αλλά δεν θα πρέπει να εμποδίζονται οι οργανισμοί αυτοί από την ε, συνεργασία τους με εμπορικές εταιρείες σε σχέση ιδιωτικού δημόσιου τομέα. Αυτός είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος να ε, διεξάγεται έρευνα σήμερα όμως δεν υπάρχει και καμία ανάγκη να παραταθεί το πεδίο της εξαίρεσης σε εμπορικές καθαρά εταιρείε, οι οποίες μπορούν να αποκτήσουν άδεια που να επιτρέπει την άντληση κειμένων και δεδομένων ώστε να έχουν την απαραίτητη νομική βεβαιότητα. Το δεύτερο θέμα το οποίο θέλω να σας υπογραμμίσω έχει να κάνει με τους εκδότες. Ε, προκειμένου να ενισχύσουμε την βιωσιμότητα αυτού του σημαντικού τομέα, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι όχι μόνο τα θέματα επιβολής καλύπτονται από την ομοθεσία μας και τις παρεμβάσεις μας, αλλά ότι ταυτόχρονα υπάρχει ένα εργαλείο ώστε οι εκδότες ε, να μπορούν να διαπραγματευτούν σωστά το θέμα της αδειοδότησης. Μπορώ ακόμη να επαναλάβω ότι η πρότασή μας ξεκαθαρίζει ότι δεν θα υπάρξει φορολόγηση των υπερδεσμών, των hyperlinks. Το τρίτο ε, θέμα έχει να κάνει με το χάσμα αξίας. Εδώ έχουμε γνώση ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια ισόρροπη αγορά εργασίας όπου οι δημιουργοί να μπορούν να εμπορεύονται τα έργα τους και να λαμβάνουν και τις σχετικές ε, απολαβές. Ε, είμαστε βέβαιοι ότι πρέπει να δημιουργηθεί εδώ κάποια ταξινόμηση. Πρώτα απ' όλα, οι κάτοχοι των δικαιωμάτων πρέπει να έχουν την ασφάλεια ότι υπάρχουν προϋποθέσεις βάσει του οποίου διανέμεται το περιεχόμενο επιγραμμικά βάσει των κανόνων για τις επιγραμμικές υπηρεσίες. Δεύτερον, να μπορούν να διαπραγματευτούν την δίκαιη αμοιβή για την ε, διανομή των έργων τους. Τρίτον, να μην περιορίζουμε τους χρήστες από το uploading και την, ε, ε, το μοίρασμα της, του περιεχομένου τους στις ανάλογες πλατφόρμες. Θα πρέπει μαζί με το Ευρωκοινοβούλιο να φροντίσουμε να υπάρξει περαιτέρω σαφήνεια για να μπορέσει η πρότασή μας να γίνει πιο στοχευμένη και πιο αποτελεσματική. Με τον κανονισμό για τα πνευματικά δικαιώματα ΣΑΠΚΑΠ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να προσφέρει ευκαιρίες στους Ευρωπαίους να έχουν ευρύτερη επιλογή για τα προγράμματα, τα τηλεοπτικά μέσω διαδικτύου στα διάφορα κρατημέλη ώστε να εποφελούνται από την πολιτιστική πολυμορφία της Ευρώπης. Η πρότασή μας σκοπό έχει να δημιουργήσει ε, τέτοιες ε, ευκαιρίες προστατεύοντας και τις αμοιβέ των κατόχων των δικαιωμάτων. Ε, διευκολύνοντας την άσκηση δικαιωμάτων για μερικούς παρόχους τηλεοπτικοακουστικών υπηρεσιών επιγραμμικά με την υποβολή, ε, με τη δυνατότητα υποβολής αίτησης ε, στο διαδίκτυο και από άλλο κράτος μέλος, προσφέρουμε περισσότερες ευκαιρίες στους παρόχους. Η πρότασή μας όμως δεν αποκλεί τη συμβασιακή ελευθερία των παρόχων και των χρηστών που θα μπορούν συμβασιακά να περιορίζουν ε, την παροχή περιεχομένου σε ορισμένες επικράτειες βάσει των εφαρμοστέων κανόνων για τα επιγραμμικά συμβόλαια. Ε, εκτιμώ τη δουλειά που έχει γίνει ως τώρα στο Ευρωκοινοβούλιο και για, τα ψηφιακά συμβόλαια και για τις δύο προτάσεις για τα ψηφιακά συμβόλαια. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων, οι συγκητές και οι βουλευτές συνέβαλαν τα μάλα Και ευχαριστώ την καθεμιά και τον καθένα σας προσωπικά για αυτό. Για το ψηφιακό περιεχόμενο και τη σχετική πρόταση, οι Υπουργοί συμφώνησαν σε μια γενική προσέγγιση στο περασμένο Συμβούλιο Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, το περασμένο Ιούνιο, και η ερχόμενη ε, Εστονική Προεδρία θα ασχοληθεί σαφώς με το θέμα αυτό για τις επιγραμμικές πωλήσει και τη σχετική πρόταση όπου η Επιτροπή Γιούρι είναι επιτροπή η οποία παρακολουθεί το θέμα. Έχουμε ήδη ξεκινήσει τις συζητήσεις στο Ευρωκοινοβούλιο, στο ε, προκαταρκτικό συμβούλιο που ετοιμάζει την Εστονική Προεδρία, αλλά και στο άτυπο ε, συμβούλιο της Εστονικής Προεδρίας τον Ιούλιο θα συζητηθούν όλα αυτά τα θέματα και η σχετική πρόταση. Οι προτάσεις για τις επιγραμμικές συμβάσεις διασυνδέεται με άλλες πρωτοβουλίες του πακέτου για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Είναι σημαντικό να το θυμόμαστε καθ' τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας. Όλα αυτά πάνε μαζί. Είναι συνδυασμένα τα ωφέλη αυτών των πρωτοβουλειών και να μην ξεχνάμε και τον απότατο σκόπο μας. Να να μεγιστοποιήσουμε τα οικονομικά κέρδη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργώντα ένα κατάλληλο περιβάλλον για τις εταιρείες και επιχειρήσεις. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να τηρούμε ε, την προσοχή μας προς το σκοπό των προτάσεων ε, για τις ψηφιακές πρωτοβουλίες να τονίσω ότι εάν θέλουμε να έχουμε χειροπιαστά αποτελέσματα για τους καταναλωτές μας και τις επιχειρήσεις μας, αυτό είναι απαραίτητο. Το μήνυμά μου προς εσάς σήμερα Είναι ξεκάθαρο και απλό. Βρέπω να υπάρχει ένα σαφή ρυθμό για την εναρμόνιση, την υψηλό επίπεδο προστασία για του καταναλωτέ με την πρόταση τη ψηφιακή αγορά υπό την Ιστονική Προεδρία, να μην τη παταλήσουμε την ευκαιρία αυτή, να μην την πετάξουμε και τέλος να ολοκληρώσω την παρέμβασή μου με λίγα λόγια για την πειρατεία. Καταλαβαίνω Μαθαίνω μάλλον ότι την τελευταία ώρα της συνεδρίασής σας ασχολήθηκατε με την πρόταση για τον ιδιωτικό βίο. Οι περισσότερες ε, αρμόδιες επιτροπές έχουν υποβάλει τα σχέδια γνωμοδότησής τους και σας ευχαριστώ για τη σκληρή σας δουλειά. Όμως στην πρόταση αυτή, ε, την δουλειά που βάλατε για την πρόταση αυτή, όμως πρέπει να πω ότι θα πρέπει να αποτιμήσουμε τις προκαταρκτικές συμφωνίες, τηρώντας το φιλόδοξο στόχο του χρονοδιαγράμματος. Βλέπουμε ότι ανακύπτουν διαφορετικές απόψεις στις κοινοβουλευτικές επιτροπές και αυτό δείχνει ότι το Κοινοβούλιο έχει μιλήσει με όλους τους ενδιαφερομένους, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι απόψεις και οπτικές γωνίες λαμβάνονται υπόψη. Παρομοίως έχουμε ε, κάνει την ανάλογη προετοιμασία για την πρόταση αυτή και πιστεύω ότι έχουμε πετύχει το σωστό σημείο ισορροπία ε, για ένα υψηλό επίπεδο προστασία του ιδιωτικού βίου, επιτρέποντα ταυτόχρονα στι εταιρείε και επιχειρήσει να έχουν καινοτομία και να αναπτύσσονται. Χωρί ε, τον ιδιωτικό βίο δεν θα υπάρχει πιστοσύνη και χωρί αυτήν οι ηλεκτρονικέ υπηρεσίε δεν θα χρησιμοποιούνται. Γι' αυτό στρεφόμαστε προς το Ευρωκοινοβούλιο και αναμένουμε την τελική έκθεση βάσει της πρότασης που θα υποβάλουμε στο τέλος του καλοκαιριού. Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε και να συνεργαστούμε μαζί σας και με το Συμβούλιο στην ανάλογη νομοθετική διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Τώρα θα απαντήσω στις ερωτήσεις σας ή θα ακούσω τις προτάσεις σας. Ελπίζω να συζητήσουμε και για το γεωγραφικό αποκλεισμό, γιατί δεν είχα πολύ χρόνο στην ομιλία μου και ήθελα να αναπτύξω και αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. you, uh, Ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε. Η κυρία Ρίγνερ ήταν η πρώτη που ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σας. Παρ' όλα αυτά έχω ένα ερώτημα. Ένα θέμα το οποίο είναι επίπεδο βεβαίω και υπάρχουν πολλές ερωτήσεις. Η δικιά μου είναι εξή. Για έναν ορισμό των ε, ψηφιακών ε, έδρων επιχειρήσεων. Ξέρουμε ότι απασχολεί βεβαίως ε, και άλλους επιτρόπους, αλλά μας αφορά εμάς και για τον υπολογισμό της ε, φορολογικής βάσης των επιχειρήσεων, γιατί διαπιστώσαμε και στα Panama Papers επιχειρήσεις που έχουν έδρες εδώ, έδρες εκεί, έδρες παραπέρα. Είναι οπωσδήποτε ένα νομικό θέμα επίσης, το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει και ακριβώς θα μιλάμε για τα ψηφιακά είναι ιδιαίτερος σημαντικό να πούμε ότι δεν έχει βρεθεί καμία λύση ή κάποιο ορισμό. Είναι οπωσδήποτε μια πρόκληση για την Κομισιόν. Οπότε το ερώτημά μου τελικά είναι το εξή. Αν η Κομισιόν σκοπεύει να ορίσει την ψηφιακή έδρα των εταιριών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Ρέντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Αντιπρόεδρε για την παρουσίαση των πολλών και σημαντικών αυτών θεμάτων. Τρία ερωτήματα έχω. Πρώτα απ' όλα συμφωνούμε όλοι ότι η ενιεύσια και η αγορά δεν μπορεί να λειτουργήσει ενώ καθένα κάνει ό,τι θέλει. Αναφέρατε τον γερμανικό νόμο περί ψευδών ειδήσεων, στον οποίο ασκήσατε μεγάλη κριτική. Και εσείς ε, και ο ειδικό Επίτροπος του ΟΗΕ για την Ελευθερία Λόγου, η δημοσιογράφοι χωρί σύνορα κτλ. Άσκησαν όλοι μεγάλη κριτική. Βλέπουμε λοιπόν από τα γερμανικά μιμιέ ότι παρόλη την κριτική ένας εκπρόσωπος της Κομισιόν ε, δήλωσε ότι καλωσορίζει την γερμανική αυτή πρόταση και πως η Κομισιόν δεν θα παρέμβει στην ε, πρόταση αυτή κατά την περίοδο ειδοποίησης. Αυτό είναι ασύνηθες γιατί η διαδικασία μετά την ε, κοινοποίηση δεν έχει οριστικοποιηθεί και τώρα ακούμε ότι η Κομισιόν δεν θα παρέμβει. Αναρωτιέμαι δηλαδή ε, τι χρήσιμότητα έχει αν δεν αγγίξουμε αυτήν την διαδικασία ε, και την οδηγία περί ηλεκτρονικού εμπορίου, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται ότι η Γερμανία μπορεί να τα αγνοεί όλα αυτά μόνο και μόνο επειδή είναι σε προεκλογική περίοδο. Θα επαληθεύσει λοιπόν την νομοθεσία αυτή η Κομισιόν και θα αναλάβει βήματα αν θεωρεί ότι δεν συμμορφώνεται με το κοινοτικό δίκαιο δεύτερον. Για την οδηγία περί copyright είπατε ότι δεν είναι αναγκαίο ή μάλλον ε, δεν είναι αναγκαίο να επεκταθεί η εξαίρεση αυτή ε, σε εταιρείε γιατί υπάρχουν άδειε διαθέσιμε στην αγορά. Δηλαδή, εγώ αν είμαι μια εταιρεία η οποία αναπτύσσω λογισμικό αναγνώριση ομιλία και χρειάζεται να επεκταθει η εξαιρεση αυτη σε εταιρειε γιατι υπαρχουν αδειε διαθεσιμες στην αγορα δηλαδη εγω αν ειμαι μια εταιρεια η οποια αναπτυσσω λογισμικο αναγνωριση ομιλιας και χρειαζεται να χρησιμοποιησω ε, εκατομμύρια εγγραφές που υπάρχουν δωρεάν στο ίντερνετ για να αναγνωρίζει έτσι την φυσική ανθρώπινη ομιλία. Πώς θα λάβω εγώ την άδεια των εκατομμυρίων ατόμων που έχουν ανεβάσει όλα αυτά τα πράγματα στο ε, διαδίκτυο. Όχι για να κάνω βεβαίως χρήση ε, των δεδομένων αυτών, Απλά για να υπάρχει η δυνατότητα να γίνει μια σύγκριση για να μάθει ο αλγόριθμος. Και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σοβαρές περιπτώσεις ε, διακριτικής μεταχείρισης με βάση τους αλγόριθμους. Π.χ. η αναγνώριση ομιλίας είναι πολύ κακή στο να αναγνωρίζει την ομιλία γυναικών, που είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Οπότε αν οι εταιρείε δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά αυτή σωστά, γιατί πρέπει να πάρουν άδειε ε, για κάτι τέτοιο, νομίζω πως ε, θα δημιουργηθεί ένα πρόβλημα. Και τέλος, για το θέμα των ε, link. Η Κομισιόν προτείνει συγγενές δικαίωμα για τους εκδότες που λέει ότι αν μεταδίδουμε μικρά κομμάτια άρθρων ε, εφημερίδων χρειάζεται μια άδεια και μετά λέει δεν ισχύει αυτό σε περιπτώσεις link που δεν απευθύνονται προς το κοινό. Δεν είναι λογικό αυτό. Δηλαδή, αν δεν απευθυνόμαστε στο κοινό, δεν χρειαζόμαστε άδεια για να απευθυνθούμε στο κοινό. Εντάξει, προφανέ. Αλλά τι γίνεται με τα αποσπάσματα άρθρων που περιλαμβάνονται στο link, στο κείμενο του URL ή συνοδεύουν το link, τον σύνδεσμο, όπως ο τίτλος ενός άρθρου. Απαιτείται έτσι άδεια για να αντιγράψουμε τον τίτλο ενός άρθρου. Στο παρελθόν ο κύριος Έτιγκερ είχε πει ότι η απάντηση είναι ναι. Σας ευχαριστώ. Και εγώ ο κύριος Άντερσον. Ευχαριστώ. Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά την συνθήκη του Μαρακές, που θα βελτιώσει την πρόσβαση στα βιβλία για άτομα με προβλήματα όρασης και ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υπερψηφίσει την υλοποίηση αυτής της συνθήκης τον επόμενο μήνα. Και αυτό με φέρνει στο επόμενο ερώτημα, που έχει να κάνει με την επικύρωση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτής της συνθήκης του Μαρακές. Αυτό πρέπει να έχει συμβεί εδώ και καιρό. Τώρα, αν αρχίσει να εφαρμόζεται, και πρέπει να ευχαριστήσω τον Επιτρόπο γιατί έχει κάνει πολύ καλή δουλειά από αυτού. Τι γίνεται με την επικύρωση λοιπόν. Για τα βιβλία. Σε αυτό το iPrint θα υπάρξει πρόταση για να αναθεώρηση οδηγία σχετικής. Κάτι έχω ακούσει Άλλοι λένε ότι δεν θα υπάρξει καμία πρόταση για να θέσει το iPrint. Υπήρξε όμω διαρροή ενό εσωτερικού εγγράφου της Κομισιόν που αναφέρεται σε κάποιες συζητήσει για την πρόταση. Δεν μπορείτε να με διαφωτίσετε. Θα υπάρξει ή δεν θα υπάρξει πρόταση για το hybrid ή ακόμα συζητείτε το θέμα. Thank you. IPRD ED is the IPR... IPRD λέτε. IPRD. Την οδηγία για την εφαρμογή, περί αυτού πρόκειται, όποιος δεν κατάλαβε. Ball. Ε, κυρία Χάνιμπολ, ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο που είναι εδώ και ε, απαντά σε ερωτήσει μας σε ό,τι αφορά την οδηγία τα πνευματικά δικαιώματα. Είναι ισορροπημένη, η πρόταση Κομισιόν την καλωσορίζω. Έχω πάντως κάποια ζητήματα που με ανησυχούν, για τις πλατφόρμες. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να παίρνουν όλο και περισσότερη εξουσία πλατφόρμες όπως το Google. Μεγάλες επιχειρήσεις που κάνουν όλο και περισσότερα και νομίζω ότι πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό και να δούμε ε, πού πρέπει να βάλουμε όρια σε αυτές τις επιχειρήσεις. Ορισμένα από αυτά που υπογραμμίσατε είναι η σωστή κατεύθυνση. Σε ό,τι αφορά τώρα την δημοσίευση, τον τύπο, είναι υποσυζήτηση, πρέπει να παραμείνει η σωστη κατευθυνση σε οτι αφορα τωρα τη δημοσιευση τον πρόταση. Το ίδιο και με το, ψηφιακό, με το αξιακό κενό. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι οι απολαβές των δημιουργών ε, και των ε, καλλιτεχνών μειώνονται σημαντικά συν το χρόνο. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε πολύ προσεκτικά με τις προτάσεις ε, που περιλαμβάνει η οδηγία. Νομίζω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Είναι λογικό, άλλωστε. Εάν υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά, πρέπει να τους στηρίξουμε, αλλιώς θα είμαστε όλοι φτωχότεροι αν πάψουν να την κάνουν. Η οδηγία είναι πολύ καλή λοιπόν και πρέπει να φροντίσουμε να κατοχυρώσουμε την ε, δίκαιη αμοιβή για καλλιτέχνες, για δημιουργούς. Επίσης, για το γεωγραφικό αποκλεισμό. Είπατε ότι ε, θέλετε να το σχολιάσετε. Σας κάνω εγώ λοιπόν την ερώτηση. πρέπει οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς είπατε να είναι ελεύθεροι, να περιορίζουν αυτά που κάνουν. Ε, μπορείτε να μας ε, πείτε κάτι παραπάνω για το γεωγραφικό αποκλεισμό και για τη χώρα προέλευσης. Εγώ πάντοτε θεωρούσα ότι το θέμα της εδαφικότητας είναι πολύ σημαντικό. Γιατί είναι και το επιχειρηματικό μοντέλο βάσει του οποίου δουλεύουν οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς και σίγουρα θα χάσουμε ποιοτικέ παραγωγές εάν αλλάξει η επικουρικότητα. Αλλά ο γεωγραφικός αποκλεισμός είναι ένα θέμα που δεν αναφέρατε και θα ήθελα να σας ακούσω γι' αυτό. Γιατί είναι και ένα σημαντικό κομμάτι των όλων αυτών ρυθμίσεων. Θα μπορούσατε ίσως λοιπόν να μας εξηγήσετε ποια είναι η θέση της Κομισιόν, η δική σας θέση για το γεωγραφικό αποκλεισμό. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ντελβό. Σύντομα παρακαλώ, γιατί μέχρι παρατέτατο θα παραμείνει ο κύριο Σάνσιπ, αν ε, δεν απατώμε. Ναι, αν το λέτε εσείς, λέει ο κύριο Σάνσιπ. I am sure he can ε, stay longer. Ε, εγώ είμαι βεβαίω ότι μπορεί να μείνει και λίγο περισσότερο. Θα είμαι πολύ σύντομη, κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα και εκτιμώ τις προσπάθειες του Επιτρόπου για την ενιαία ψηφιακή αγορά. Και βλέπω ότι υπάρχουν δυσκολίες και μεγάλη αντίσταση από πολλά κράτη-μέλη για αλλαγή της νομοθεσίας. Άρα, ο σωστός τρόπος είναι να υιοθετηθεί κοινή νομοθεσία πριν υιοθετήσουν δική του νομοθεσία τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό λοιπόν και συντάξαμε την έκθεσή μας για τη ρομποτική και τις νομικές επιπτώσεις που έχει η ρομποτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να πω ότι με απογοήτευσε ιδιαίτερα η αντίδραση της Κομισιόν που ναι μεν συμφώνησε με την ανάλυση μας αλλά δεν προέβησε καμιά συγκεκριμένη πρόταση. Σας παρακαλώ λοιπόν, ιδίω ότι αφορά την ευθύνη. Θα έχουμε αυτά τα οχήματα χωρίς ε, οδηγό στους δρόμους και στη Γερμανία ήδη γίνονται κάποιες προσπάθειες για την κατάρτιση ενός νομοσχεδίου για την αστικευτή. Αν έχουμε εναρμόνιση πριν υιοθετήσει το κάθε μέρο τη δική του νομοθεσία, θα προλάβουμε, αλλιώς θα τρέχουμε σε τις εξελίξεις. Ας έχουμε λοιπόν έστω και μια χτίδα ελπίδα ότι μπορεί η Κομισιόν να καταθέσει μια πρόταση για την ευθύνη πριν τα τέλη του έτους. Ισχύει αυτό ή όχι, κύριος Φως. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το λόγο και που ήρθατε. Πρώτα απ' όλα το θέμα και το έθεσα και στον κύριο Τίμερμανς έχουμε συγκεκριμένα νομοθετήματα που συνδέονται είτε πλευρά ουσία είτε εξορισμού. Η privacy, κώδικα επικοινωνιών, ο κώδικα επικοινωνιών με το ψηφιακό περιεχόμενο. Και έχω την εντύπωση ότι έχουμε διαφορετικές ε, υπηρεσίες κομισιών που δεν συνεννοούνται. Το ερώτημα είναι λοιπόν πώς θα διασφαλίσουμε σε όλον αυτόν τον ψηφιακό τομέα ότι θα υπάρχει ένα ενιαίο δίκαιο. Γιατί είναι δύσκολο. Φαίνονται όλα αυτά κάπως ε, ασύνδετα. και βλέπουμε ότι το ένα νομοθέτημα εδώ πέρα υπονομεύει το άλλο. Και το τι γίνεται με το 5G. εδώ πέρα θα πρέπει να σκεφτόμαστε θα έλεγα σε gigabyte, όχι σε megabyte για το τι θα προκύψει σε upload, download κτλ. Και βεβαίω όσον αφορά το ψηφιακό περιεχόμενο υπάρχουν και τα δύο ουσιαστικά ερωτήματα. Το ένα, η σχέση με την οδηγία προστασίας δεδομένων και το άλλο είναι ως δεδομένα ως αντιστάθμισμα. Είναι αυτό λογική για να διατηρήσουμε την ιδιωτική σφαίρα. Και το άλλο μου ερώτημα είναι ε, το ότι θέλουμε να ρυθμίσουμε ακριβώς την ιδιοκτησία των δεδομένων. Ειλικρινά θα μπλέξουμε και δεν θα μπορέσουμε να βγούμε ποτέ αν αρχίσουμε να ψάχνουμε ποιος έχει ποια δεδομένα και πότε. Το θέμα της ιδιοκτησίας των δεδομένων δεν θα μας ε, οδηγήσει πουθενά. Θα πρέπει βεβαίως ακριβώς να δούμε πως ε, θα τα ξεβλέξουμε και στο μυαλό μας κάποια στιγμή. Θα πρέπει δηλαδή να δούμε διαφορετικά τελείως το ψηφιακό πεδίο με θάρρος, με δημιουργικότητα, γιατί με την ε, παλιά νοοτροπία δεν θα μπορέσουμε να το συλλάβουμε. Σας ευχαριστώ. Ähm, ναι, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να αναφερθώ στο ερώτημα της κυρίας Χάνιμπολ για, το... για τον γεωαποκλεισμό. Μπορείτε να μας πείτε κάτι για το τι γίνεται με την περίπτωση του Sky. Και να δούμε το πώς ε, μπορεί να επηρεάσει τον ε, γεωαποκλεισμό. Και πώς θα μπορούσε να είναι αδύνατος κάτι τέτοιο στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Πόσο λεπτά. Πόσα λεπτά. Με το πάσο σας, λέει ο πρόεδρος. μα τι θα πει με το πάσο μου δηλαδή. Ε, θα πει, απαντήστε, αλλά σύντομα, αλλά ικανοποιήστε και όλους τους βουλευτές. Μάλιστα, μάλιστα. Ε, δύσκολα, δύσκολα μου βάζετε. Λοιπόν, τους φόρους. Λοιπόν, είπαμε ότι οι φόροι πρέπει να καταβάλλονται στις χώρες ε, όπου δημιουργείται το κέρδος. Και το θέμα αφορούσε τον ε, ορισμό της ε, ψηφιακής επιχειρηματικότητας και βεβαίως ε, όταν λέμε, λέμε ότι πρέπει να πληρώνουν φόρους εκεί όπου δημιουργείται το κέρδος ε, πρέπει να εξηγήσουμε και τι σημαίνει αυτό αλλά εγώ δεν έχω κάποιον έτοιμο ορισμό μετά για το γερμανικό αυτό νόμο είναι λίγο νωρίς για να σχολιάσουμε αλλά Φαίνεται ότι, ναι, κοινοποίησαν αυτόν τον νόμο, το σχέδιο νόμου και είχα και κάποιες συζητήσεις ε, με τον Υπουργό και ε, από ό,τι καταλαβαίνω έγιναν κάποιες διορθώσεις ήδη ε, κάποιες διορθώσεις εκεί όπου υπήρχαν κάποια νομικά ζητήματα εκεί όπου υπήρχαν κάποιες υποχρεώσεις κοινοποίησης ε, σύμφωνα με το γερμανικό νόμο. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια νομικά ζητήματα, αλλά δεν ανησυχώ τόσο για τη Γερμανία. Η εφαρμογή του νόμου αυτού στην Γερμανία οπωσδήποτε θα είναι τέλεια, αλλά το τι θα γίνει σε άλλα κράτη-μέλη δεν το ξέρω. Ε, εγώ είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει κάποια κατάχρηση άρθρων και παραγράφων ε, του νόμου αυτού. Το τι θα γίνει σε άλλες χώρες που θα ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτού του νόμου και ξέρουμε όλοι ποιες χώρες εννοώ. Έχω κάποιες ε, σοβαρές επιφυλάξεις και δεν είμαι έτοιμος να πω πώς θα δράσει η Κομισιόν. Είχαμε χρόνο να αποφασίσουμε και εάν δεν καταλήξουμε σε κάποια γνωμοδότηση ε, και κάποια γνώμη ε, επιφυλασσόμαστε. Θα δούμε λοιπόν αν κάποια άρθρα είναι αντίθετα με το ευρωπαϊκό δικαίωμα, οπωσδήποτε θα παρεμβούμε. Τώρα για την ε, συλλογή δεδομένων, όπως είπα, και κειμένου. Όπως είπα πολλές φορές, το θέμα δεν είναι η συλλογή κειμένου και δεδομένων, αλλά αφορά το ότι πρέπει να έχουμε την ίδια προσέγγιση σε όλα τα θέματα. Κοιτάμε και την πολιτική πραγματικότητα, τι είναι εφικτό και τι δεν είναι εφικτό. Οπότε η πρότασή μας σε ήταν και ακόμα πιο φιλελεύθερη από τις πιο φιλελεύθερες λύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι η Βρετανική προσέγγιση. Οπότε δεν νομίζω ότι πρέπει να καταστρέψουμε κανένα επιχειρηματικό μοντέλο που λειτουργεί σήμερα. Ταυτόχρονα όμως γνωρίζουμε ότι η συλλογή κειμένων και δεδομένων στα περισσότερα κράτη-μέλη δεν ε, υπάρχει ως δυνατότητα για τους επιστήμονες. Ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μια πρωτοπορία, αλλά πρόκειται κυρίως για επιστημονικά άρθρα που δημοσιεύονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε για τα μικρότερα κράτη-μέλη ε, δεν, να, δεν υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες για τους επιστήμονες. Νομίζω λοιπόν ότι η πρότασή μας ήταν πολύ ισορροπημένη. Και δεν ε, θα ήθελα τώρα να ε, ξεκινήσω την πιο φιλόδοξη πρόταση στον κόσμο που θα κρατήσει δεκαετίες, θα συζητείτε δεκαετίες χωρίς αποτέλεσμα. Εγώ θα ήθελα κάποια αποτελέσματα. Γι' αυτό ακριβώς εξετάζουμε και γνωμοδοτήσει σε διαφορετικά κράτη-μέλη, στο κοινοβούλιο, σε διάφορε επιτροπέ κτλ. Θα προφυλάξω λοιπόν την σχετική πρόταση του copyright, αλλά είμαι όπως εδώ ήταν εκτός καλές ιδέες για το πώς μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερη πρόταση για τους συνδέσμους. Όπως σωστά αναφέρεται, Το κείμενο αναφέρει ότι τα συγγενή δικαιώματα για τους εκδότες δεν σημαίνουν ότι θα απαγορευθούν ή θα φορολογηθούν ε, οι σύνδεσμοι. Όταν μιλάμε για συνδέσμους, ε, το περιεχόμενο αυτό ήδη προστατεύεται από το copyright γιατί οι κατοχή των δικαιωμάτων είναι δημοσιογράφοι, φωτογράφοι. Και θα, ε, εντάξει, και θα, θα συμμορφωθούν οι εκδότες. Εντάξει, μπορείτε να διαφωνείτε, αλλά είμαι πεπισμένος ότι η πρόταση αυτή ήταν πολύ ισορροπημένη και για να είμαι ειλικρινής δεν ε, μπορώ να δω κάποιον ε, λόγο για να ξανανοίξει η πολύ καλή νομολογία που έχουμε για τους συνδέσμους και υπερσυνδέσμους ε, που έχουμε με την εισηγήτρια την κυρία Κομοντίνη. Είχατε κι εσείς ε, συζητήσει αυτά τα ζητήματα και μάλλον θα συνεχίσουν αυτές οι συζητήσεις στο Κοινοβούλιο. Ε, το είχα πει και πέρσι, ήταν κρίμα το ότι χρειάστηκαν τόσα χρόνια ε, για να διορθωθεί αυτή η συνθήκη. Τέλος ε, για την κύρωση αυτής της διαδικασίας. Νομίζω ότι είναι ένα βήμα προς την ε, σωστή κατεύθυνση. Και πάλι πρέπει να δούμε τα άτομα με αναπηρία, τους τυφλούς, να έχουν πρόσβαση. Οπότε Αυτές οι διοργανικές ε, συζητήσεις είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί. Έχουμε βεβαίως και το 10 και ελπίζω σύντομα να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Τέλος. για την οδηγία περί επιβολής ε, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Θα επανεξετάσουμε αυτήν την οδηγία και θα υποβάλουμε τις προτάσεις μας, αλλά πρέπει να πω ότι θα χρειαστεί λίγος χρόνος. Πρώτα απ' όλα, θα θέλαμε να ε, δούμε αυτές τις λύσεις αυτορύθμισης. Ε, την αρχή ακολουθούμε το χρήμα Και υπάρχουν και πέντε διαφορετικά παραδείγματα συνεργασίας για να δούμε τις μεταφορές, την διαφήμιση κτλ. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ καλύτερη η εθελοντική λύση, η αυτορύθμιση, παρά κάτι το αυστηρότερο το οποίο θα προσπαθήσει να ρυθμίσει οριζοντίως όλα αυτά τα ζητήματα. για όλες αυτές τις περιπτώσεις ε, παραβιάσεων. Για το πλαφόν, ε, πράγματι, είναι ένα πρόβλημα όχι περισσότερο για τον απλό κόσμο, αλλά π.χ. για τους μουσικούς. Έχουμε διαφορετικές πλατφόρμες, άλλες πλατφόρμες βασίζονται σε συνδρομή, έχουν ε, π.χ. 140 εκατομμύρια συνδρομητές κάθε μήνα και δίνουν 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε μουσικούς. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν άλλες πλατφόρμες που βασίζονται σε διαφημίσεις ε, που έχουν κοντά στο 1 δισεκατομμύριο επαφές ανά μήνα αλλά στους μουσικούς δίνουν 0,6 ε, δισεκατομμύρια ευρώ. Και βεβαίω αντιλαμβάνομαι τους μουσικούς που λένε ότι υπάρχει ένα χάσμα στην αξία. Και βεβαίως ε, υπάρχει και το θέμα ακριβώ του ψηφιακού περιεχομένου. Η πρόταση είναι πολύ ισορροπημένη θα έλεγα. και δεν αντιβαίνει την οδηγία περί ηλεκτρονικού εμπορίου. τι γίνεται με τους ιδιοκτήτες των δικαιωμάτων και την αμοιβή τους, γιατί σήμερα οι δημιουργοί δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι. Η ταυτοποίηση του περιεχομένου βεβαίως δεν είναι τόσο ακριβή όσο νομίζει ο κόσμος. Πάντα δίνουν το παράδειγμα του YouTube που το έχει ξεκινήσει από το 2007 και λένε ότι επένδυσαν 60 εκατομμύρια δολάρια για να βρουν αυτή τη λύση. Αλλά υπάρχουν ε, και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών, το Audible παραδείγματο χάρη, που μπορεί να ταυτοποιήσει 10.000 τραγούδια και γι' αυτό πλήρωσαν 500-600 δολάρια. Ε, και 90% των ερωτηθέντων ε, επί του θέματος ε, είπαν ότι θα θέλαμε να έχουμε κάποια αμοιβή για το περιεχόμενο, ενώ οι υπόλοιποι λένε κατεβάστε το. It's Uh, είναι μεγάλο το θέμα για τους μουσικούς. Και είναι άδικο το να συνεχίσουμε όπως κάνουμε. Για τα ζητήματα αστικής ευθύνης. Είχαμε την οικονομία των δεδομένων ε, στο σύνολό της και πρέπει να μιλήσουμε για τις ε, ροές δεδομένων, τις ελεύθερες ροές, που απαιτούνται οπωσδήποτε για την οικονομία των δεδομένων, αλλά πρέπει να δούμε επίσης ε, και τα ζητήματα τα καινούργια, όπως παραδείγματος χάρη ναι, τα ζητήματα αυτά ευθύνης δεδομένων. Θεωρώ λοιπόν ότι θα είμαστε έτοιμοι τον Σεπτέμβριο να καταθέσουμε την πρότασή μας για αυτό το θέμα και δεν είμαι τώρα τόσο αισιόδοξο, δεν μπορώ να πω ότι θα γίνει φέτος γιατί ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι πρακτικές διαφέρουν και δεν θέλω να πω τώρα ότι κάποιες είναι καλές και κακές. Παραδείγματος χάρη, Οι Siemens, η σκάνια δεν θέλουν να έχουν τα δεδομένα στην ιδιοκτησία τους, θέλουν πρόσβαση λένε. Και λένε όσοι έχουν τα φορτηγά θα έχουν και την ιδιοκτησία των δεδομένων. Η TomTom ταυτόχρονα θέλει την ιδιοκτησία των δεδομένων και τι μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι μια πρακτική είναι καλή, πώς μπορούμε να πούμε ότι μια πρακτική είναι καλή και η άλλη όχι. Με την ευθύνη λοιπόν είναι δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να αλλάξουμε τις προτάσεις μας. Αλλά δεν είμαι έτοιμος αυτή τη στιγμή να πω πώς ακριβώς. Για τον κανονισμό περί ηλεκτρονικής ιδιωτικότητας και προστασίας των δεδομένων. Δεν νομίζω ότι αρκεί ε, να έχουμε έναν γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων δεν θα καλύπτει όλους αυτούς τους προβληματικούς τομείς που θα θέλαμε να καλύπτει. Αλλά όταν ξεκίνησε αυτή η πρόταση κανονισμού, στόχος μας ήταν αρχικά να εναρμονίσουμε αυτούς τους κανόνες ε, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί σήμερα έχουμε την οδηγία τη σχετική, αλλά η εφαρμογή της βεβαίως διαφέρει από χώρα σε χώρα. Οπότε θα θέλαμε να αναγνωρίσουμε αυτούς τους κανόνες. Μετά θέλουμε να δημιουργηθούν και οι ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ τηλεπικοινωνιακών εταιριών και των άλλων εταιριών που είναι over the top. Ε, βεβαίω αυτό σημαίνει ότι ε, εμπιστευτικέ είναι μόνο όταν μιλάμε για εταιρείε τηλεπικοινωνιών. Και βεβαίω δεν είχαμε σοβαρά προβλήματα και με τις άλλες ε, εταιρείε, αλλά νομικά μιλώντας δεν καλύπτονται. Και σύμφωνα με την δημόσια διαβούλευσή μας, ο κόσμος θα ήθελε νομικά μιλώντας να προστατεύεται ε, δια νόμου η εμπιστευτικότητά τους. Μιλάμε για πολύ ψηλά ποσοστά, από 80-90% λοιπά. Δεν είναι δηλαδή 50-50 ας πούμε. Οπότε, Η εμπιστευτικότητα οπωσδήποτε είναι πάρα πολύ σημαντική και αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν ε, κάποια ζητήματα που αφορούν ε, τις διαδικασίες, ε, κυρίως τι επιλογές έχουμε για τα cookies Ο κόσμος δεν θέλει κάτι τέτοιο. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι πάλι θέλουν να υπάρχει ιδιωτικότητα από τον σχεδιασμό ήδη. Άλλοι λένε ότι ο κανονισμός αυτός δεν χρειάζεται καθόλου. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι η πρότασή μας εξακολουθεί να είναι ισορροπημένη αλλά από αυτού του ζητήματο η Κομισιόν είναι ανοιχτή για να ακούσει όλου του ενδιαφερόμενου. Μετά. Για το γεωγραφικό αποκλεισμό. Όπως είχα πει ξανά και ξανά, η αρχή της εδαφικότητας είναι πολύ σημαντική και για τη δική σας την Επιτροπή, διότι πρέπει να προστατευτεί. Ωστόσο, έπρεπε να, προβλέψουμε, να και την άμυνη πρόσβαση για το ψηφιακό περιεχόμενο των πολιτών σήμερα. Οι άνθρωποι που επιθετικά ε, προστατεύουν την εδαφική τους αποκλειστικότητα, ε, με κάθε τίμημα δεν δίνουν καμία σημασία στην ε, μια κάποια παραβίαση. Το 20% των χρηστών του διαδικτύου στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιούν τις διευθύνσεις, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις IPN για, και τις αλλάζουν για να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο παλού. Δεν είναι δύσκολο να αλλάξει κανείς ε, τη διεύθυνσή του και να χρησιμοποιήσει το VPN ε, με κάτι σαν 20 ευρώ το μήνα. Και ο κόσμος δεν σκέφτεται ότι κάνει κάτι κακό. Αλλά εδώ υπάρχει πρόβλημα. Διότι δεν πάνε οι αμοιβέ εκεί που πρέπει. 68% των ε, θεατών ταινιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση λένε ότι χρησιμοποιούν τα δωρεάν download. Τι θα πει δωρεάν κατέβασμα. Θα πει δωρεάν περιεχόμενο και κατά καιρού, από καιρού καιρών υπάρχουν κάτι επιπλοκέ, αλλά ο κόσμο τα αντιμετωπίζει. Και πάλι υπάρχει πρόβλημα για του δημιουργού. Δεν παίρνουν την αμοιβή που του αναλογεί. Η δική μου λοιπόν η κατανόηση για την απόλυτη αποκλειστικότητα είναι απλή ή 0 ή 100% αλλά απόλυτη αποκλειστικότητα δεν γίνεται. Κάτι μεταξύ του 0 ή του 100. Δεν το καταλαβαίνω. Ενώ στην πραγματική ζωή φτάνει από το 20-68% αυτή η απόλυτη αποκλειστικότητα. Να αναγνωρίζουν όλοι, ακόμη και οι παραγωγοί, που πουλάνε και διαφημίζουν αυτή την αποκλειστική εδαφικότητα σε κάποιους. Δεν υπάρχει και δεν γίνεται στην πραγματική ζωή. Οπότε... Έπρεπε να βρούμε κάποια συμφωνία σε σχέση με την πρόταση για το γεωγραφικό αποκλεισμό, μιλώ για τον αδικαιολόγητο γεωγραφικό αποκλεισμό και για άλλη μια φορά πήγαμε με την προσέγγιση βήμα προς βήμα. Ήδη με την κατάρριξη των τελών περιαγωγής, την φορητότητα, και την κατάργηση του γεωγραφικού αποκλεισμού θα υπάρξει πρόοδος για τους πολίτες. Το περιμένουν πώς και τι. Το αναμένουν και καραδοκούν. Θα σας παρακαλέσω να είστε κι εσείς λοιπόν επικοδομητικοί σε όλες αυτές τις συζητήσεις, αλλά ταυτόχρονα να συνεργαστούμε. Το σκαί υπόθεση με πολιτικό χαρακτήρα. Ξέρουμε ότι αυτές οι υποθέσεις είναι πολύ συγκεκριμένε. Είναι πολύ συγκεκριμένε πληροφορίες που αφορούν μια πολύ συγκεκριμένη εταιρεία. Δεν μπορεί κανείς να προβλέψει τι θα γίνει με την Sky Είναι όλες τις άλλες εταιρείες. Διότι οι καταστάσεις αυτές είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους και δεν μπορεί κανείς να τα βάλει όλα στο ίδιο σακούλι. και για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να λειτουργήσει ως copy-paste στην περίπτωση αυτή και να βρεθεί λύση για όλες τις ανάλογες περιπτώσεις. Είναι θέμα εφαρμογής της οδηγίας. Σας ευχαριστώ. Και εμείς πολύ σας ευχαριστούμε, Αντιπρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ για όλες τις απαντήσεις με τις οποίες καλύψατε τις σημερινές ερωτήσεις. Καταλαβαίνω ότι θα μπορούσατε να μείνετε ώρες εδώ και να συζητάμε, διότι τα θέματα που αντιμετωπίσατε είναι ευρύτατα. Ελπίζω ότι στα πλαίσια του διαρθρωμένου διαλόγου θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας και αναμένω την ερχόμενη συνεδρίαση μαζί σας.